Uh, good afternoon, everybody. Uh, welcome to the... Καλησπέρα σας. Uh, καλώς ήρθατε στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Θα ξεκινήσουμε ένα δεύτερο σημαντικό θέμα σήμερα το, φακε... του... σήμερα το απόγευμα για την έγκριση τύπου των ε, δίτροχων και τρίτροχων ε, ε, οχημάτων. Καλωσορίζω τον εισηγητή και τον κύριο Ματίνο από την DG Enterprise DG Επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ που καθίσατε και το απόγευμα, ήσασταν μαζί και το πρωί. Σας κρατήσαμε απασχολημένοι στο Κοινοβούλιο όλη μέρα. Ποιος άλλος είναι εδώ? Η Αντιπρόεδρος, ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ε, που είναι και σκιώδης ηγητής για την ομάδα Γκουε. Και εγώ θα είμαι σκιώδης ηγητής για τη δική μου ομάδα. Οι πράσινοι, οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλιστές ε, θα ακούσουν τους σκιώδεις τους σε ευθέτω χρόνο. Τώρα καλό είναι να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Και όσοι ήθιστε, στην Επιτροπή μας θα ακούσουμε μια παρουσίαση της, αξιολόγησης, ε, της μελέτης αξιολόγησης της ε, Επιτροπής για να καταλάβουμε το θέμα και μετά θα μας κάνει μια παρουσίαση και ο εισηγητής. Πρώτα η Κομισιόν και μετά ο εισηγητής βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές διαφάνειες. Όσοι μας βλέπουν από το ίντερνετ έχουμε τις διαφάνειες. Δύο ειδών διαφάνειες. Και αν κάποιος ε, μας παρακολουθεί μέσω του ίντερνετ ε, και ενδιαφέρεται να λάβει αντίτυπα, μπορεί η γραμματεία μας να σας στείλει. Επίσης, μπορείτε να υπογράψετε το newsletter της Επιτροπής ΕΜΚΟ ε, είναι best seller τώρα. Ε, χίλια άτομα έχουν υπογράψει στο ίντερνετ ε, αυτό το newsletter. Είμαστε η πρώτη επιτροπή που σπάσαμε το όριο των χιλίων υπογραφών. E Στην η διεύθυνση. Το κοινό λοιπόν, αν ενδιαφέρεται, άκουσε τα στοιχεία. Τελειώσαν οι διαφημίσεις για σήμερα το απόγευμα και τώρα ο κύριος Ματίνο, Τζάκομο Ματίνο, θα παρουσιάσει την μελέτη αντικτύπου σε αυτή την τόσο σημαντική πρόταση για τα δίτροχα, τρίτροχα και τετράτροχα οχήματα. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους πάντες. Σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια και την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα το πρωί μετά τα τρακτέρ ε, που παρουσιάσαμε, να παρουσιάσουμε τα οχήματα της κατηγορίας L, ε, δίκυκλα και μοτοποδήλατα κτλ. Ελπίζω να μην σας ε, ενοχλήσω με κάποιες αναφορές, με κάποιες έννοιες. Σήμερα το πρωί κάναμε κάποια γενικά σχόλια. Καλό είναι να παρουσιάσουμε το γενικό πλαίσιο. για να ακούσουμε και να ε, καταλήξουμε σε μία ε, σφαιρική θεώρηση για το σύστημα έγκρισης τύπου για τα επιβατικά αυτοκίνητα. Είχαμε κάνει μια πρόταση. Σήμερα το πρωί ακούσαμε την παρουσίαση της μελέτης αντικτύπου για τα γεωργικά και οχήματα και τα τρακτέρ και τώρα πάμε στα... στην κατηγορία L. Ο στόχος είναι η απλούστευση και η καλύτερη νομοθεσία να μην ξεχνάμε τους στρατηγικούς ε, προσανατολισμούς της ομάδας υψηλού επίπεδου ΚΑΣ 21 ε, που τώρα δεν ε, υπάρχει πια. Εδώ και ένα μήνα έχουμε μια νέα ομάδα υψηλού επίπεδου. Το πλαίσιο είναι ο εξορθολογισμός του νομικού συστήματος. Να σας μιλήσω για μια διαφορά με, την πρόταση για τα γεωργικά και δασοκομικά οχήματα. Σε αυτή την περίπτωση η Κομισιόν θεωρεί ότι είναι πολύ χρήσιμο να επικαιροποιήσουμε τις απαιτήσει για την ασφάλεια, για το περιβάλλον και ένα νέο στοιχείο για την νομοθεσία έγκρισης τύπου, να έχουμε και διατάξεις για την εποπτεία της αγοράς. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια να υπενθυμίσω σύντομα τι περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογή της πρότασης. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι ότι έχουμε μια τεράστια κατηγορία, πολλά προϊόντα, πολύμορφα. Ξεκινάμε από κάποια οχήματα ηλεκτρικά ε, ποδήλατα δηλαδή συγκεκριμένης ισχύω μέχρι τα μίνι αυτοκίνητα όπως λέμε ή παρόμοια οχήματα, δηλαδή τετράτροχα, παντός εδάφου, ε, για το δρόμο, οχήματα για το δρόμο και μοτοσυκλέτες από μοτοποδήλατα, μοτοποδήλατα δηλαδή μέχρι καλές μηχανές, νατές μηχανές. Λοιπόν, τα θέματα τα οποία καλύπτει η μελέτη αντικτύπου πολύ σύντομα. Κλασικό θέμα στην έγκριση τύπου είναι το περίπλοκο του πλαισίου. Ο στόχος είναι απλούστευση και εξορθολογισμός λοιπόν της νομοθεσίας. Όταν εξετάζουμε τις εκπομπές, το επίπεδο των εκπομπών αυτού του κλάδου αν κοιτάξουμε τις συνολικές εκπομπές των οδικών μεταφορών, είναι αρκετά σημαντικός, παραμένει σημαντικός παρότι υπάρχει μια συνολική πτωτική τάση των εκπομπών από τις οδικές μεταφορές. Σε αυτό το τομέα λοιπόν έχουμε επίσης μια ε, ανησυχία ε, τι θα γίνει με το θέμα της ασφάλειας. Θα μπω και σε λεπτομέρειες για το θέμα της ασφάλειας σε λίγο. Για τις νέες τεχνολογίες, επίσης, το σημερινό νομικό πλαίσιο δεν είναι ιδανικό και αυτό είναι ένα θέμα, μια πρόκληση για όλη την νομοθεσία έγκρισης τύπου. Για τα μοτοποδήλατα και τις μηχανές ε, είναι πολύ πιο έντονο το πρόβλημα από ό,τι για άλλα προϊόντα. Είναι ένας τομέας ο οποίος είναι προφανώς πολύ καινοτόμο και το να εξασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα που εμπεριέχουν νέα τεχνολογία μπορούν να τεθούν γρήγορα στην αγορά, στο βαθμό που πληρούν τις συνολικές απαιτήσεις. Θεωρούμε ότι είναι σημαντική ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν βάλαμε και αυτό το σημείο στην, στα προπασκευαστικά στάδια, δηλαδή ε, δημόσια συζήτηση, διαβούλευση και μελέτη αντικτύπου. Όπως σας είπα στην αρχή, το θέμα της εποπτείας της αγοράς είναι κοινό σε όλες τις ε, νομοθεσίες έγκρισης τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση των τρακτέρ, ε, το χρονοδιάγραμμα δεν μας επέτρεψε να ενσωματώσουμε κάποιες από τις διατάξεις, διότι η οριζόντια νομοθεσία, ή το νέο νομοθετικό πλαίσιο όπως λέγεται, δεν είχε ολοκληρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση όμως, με περηφάνεια σας ανακοινώνουμε ότι εργαστήκαμε πολύ σκληρά, ούτως ώστε να ενσωματώσουμε με συνέπεια ελπίζω τις διατάξεις ε, του νέου νομοθετικού πλαισίου σε αυτή την νομοθετική πρόταση. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι για τα οχήματα της κατηγορίας L κάτι που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι οι αρχές και οι καταναλωτές σημειώνουν ότι Υπάρχουν πολλά προϊόντα τα οποία δεν συμμορφώνονται ή συμμορφώνονται οριακά με τις προϋποθέσεις έγκρισης τύπου και αυτά τα προϊόντα μπαίνουν στην αγορά. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα στα πλαίσια αυτής τη πρότασης. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Η νομική διάρθρωση και το θέμα της απλούστευσης. Πολύ σημαντικό. Όπως ε, και σε άλλες προτάσεις και εδώ προτείνουμε ένα κανονισμό, ε, μια πράξη συναπόφασης που θα συνδυαστεί με πράξεις ε, κατεξουσιοδότηση καθώς και τις εφαρμοστικές πράξεις που αφορούν τα διοικητικά και διαχειριστικά θέματα. Σε αυτή την περίπτωση προτείνουμε να μπούμε σε εξυγχρονισμό των τεχνικών προϋποθέσεων, επικαιροποίηση των τεχνικών προϋποθέσεων, που είναι πολύ σημαντικό για να πετύχουμε και σε επίπεδο ποιότητας και σε επίπεδο χρόνου ε, ικανοποιητική ολοκλήρωση των εφαρμοστικών μέτρων και των ε, πράξεων κατεξουσιοδότηση. Δηλαδή, θα έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση σε πακέτο μία πράξη εξουσιοδότηση που θα αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα και τα θέματα των επιδόσεων και μία ακόμα για τα θέματα της ασφάλειας. Και μία τρίτη ε, προϋποθέσεις για την κατασκευή των οχημάτων. Τώρα θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες για τα στοιχεία της ε, μελέτης ε, αντικτύπου ό,τι αφορά την ασφάλεια. Το πρώτο σημείο το οποίο πρέπει να εξετάσουμε είναι οι στατιστικές που αφορούν τα μοιραία τροχαία ατυχήματα και τους σοβαρούς τραυματισμούς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει μεγάλη σημασία στη βελτίωση της ασφάλειας των δρόμων μας στην Ευρώπη αν προσπαθήσουμε να διαχωρίσουμε, και να εντοπίσουμε την κατηγορία L, δηλαδή μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα, βλέπουμε ότι αναλογικά, δυστυχώς, αυτός ο τομέας ε, παρουσιάζει μεγάλο αριθμό και ποσοστό ε, και μοιραίων τροχαίων αλλά και σοβαρών ε, ατυχημάτων. Επίσης σημαντικό είναι ότι όταν κοιτάζουμε τα στοιχεία, άλλα, άλλοι τρόποι μεταφοράς με οχήματα ε, παρουσιάζουν μείωση και στα ατυχήματα και στους θανάτους. Δυστυχώς τα οχήματα της κατηγορίας L δεν παρουσιάζουν αυτή την μείωση. Για να μην πω υπάρχει και μια ελαφρά αύξηση στα νούμερα και κατά απόλυτο τιμή και σε επίπεδο ποσοστού. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο η Κομισιό με την πρότασή της θέλει να αντιμετωπίσει. Θέλουμε να πετύχουμε ένα ικανοποιητικό στόχο, ούτως ώστε μέσω, μέσω της έγκρισης τύπου να συνεισφέρουμε στη μείωση των ατυχημάτων και στην αύξηση της ασφάλειας των ευρωπαϊκών δρόμων. Κάτι το οποίο βεβαίως εξαρτάται και από πολλούς άλλους παράγοντες, αλλά και εμείς θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να συμβάλλουμε όσο μπορούμε ούτως ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή έγκριση τύπου και τα καλύτερα δυνατά τεχνικά χαρακτηριστικά. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ποια είναι τα θέματα που διακυβεύονται μέσω της μελέτης αντικτύπου. Αποφυγή των ατυχημάτων, καταρχάς. Όταν τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να παίξουν ένα ρόλο, να παίξουν. Και μετριασμός των τραυματισμών σε περίπτωση ατυχημάτων. Επομένως προστασία πριν και όταν γίνεται μετά το ατύχημα. Επόμενη διαφάνεια. Οι εναλλακτικέ λύσεις που εξετάσαμε είναι κοινή πρακτική της μελέτης αντικτύπου. Δεν προβλέπουμε αλλαγή στις τρέχουσες προϋποθέσεις. Αυτή ήταν η μία επιλογή. Η άλλη επιλογή ήταν υποχρεωτική εισαγωγή του ABS σε όλα τα δίτροχα. Επίσης, διαβάθμιση των μέτρων για τα πιο, τους πιο ισχυρούς κινητήρες να έχουμε ABS ενώ για τα λιγότερο, τις λιγότερο ισχυρές μηχανές και κινητήρες τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και άλλες τεχνολογίες όπως παραδείγματο χάρη συνδυασμό ε, μέσων τροχοπέδησης. Τέλος, η άλλη εναλλακτική λύση. Σημειώνουμε, πρέπει να σημειώσουμε, ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία κατασκευαστών ε, μηχανών, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών. Από το 2004 ε, εθελοντικά δεσμεύεται να προσφέρει το σύστημα του ABS ή ένα συνδυασμένο σύστημα τροχοπέδησης στα μοντέλα της. Επομένως υπάρχει μια εθελοντική δέσμευση από τον κλάδο και αυτό αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο τμήμα της ευρωπαϊκής αγοράς, αλλά δεν καλύπτει όλους τους κατασκευαστές, πρώτον, αυτό είναι το ένα πρόβλημα, και δεύτερον, αυτή η αυτοδέσμευση, αυτή η εθελοντική δέσμευση, καλύπτει προαιρετικά, υπάρχει μια προσφορά αυτών των συστημάτων και ο πελάτης, ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα ανάλογα με την τιμή που θέλει να πληρώσει για το προϊόν, το, προϊόν, το τελικό προϊόν, να αγοράσει ή όχι αυτό που προσφέρουν οι κατασκευαστές. Επόμενη διαφάνεια. Η μελέτη αντικτυπίου η μελετη αντικτυπιου μιλαει και για θέματα και για μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας. Η βασική ανησυχία εδώ είναι ότι κατά το τιμή Αν συγκρίνουμε με τα ελαφρά εμπορικά οχήματα και με τα επιβατικά οχήματα, ε, τα νούμερα δείχνουν κάτι ανησυχητικό. Υψηλό μερίδιο εκπομπών ε, υδρογονανθράκων, διοξιδίου του άνθρακα και σωματιδιακή ύλη. Ε, σωματιδιακής ύλης. Βλέπετε ότι μέχρι το 2020 αν δούμε το μερίδιο που θα εκπέμπεται από τα οχήματα αυτά της κατηγορίας L, σε συνδυασμό, σε σύγκριση μάλλον, με όλες τις εκπομπές υδροκονανθράκων παντός εδάφους, αυτό το ποσοστό της κατηγορίας L αυξάνεται. Και βεβαίως αυτό θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε με νομοθετικά μέσα. και έχουμε κάνει και διάφορες μελέτες. Η επόμενη διαφάνεια παρουσιάζει τα προβλεπόμενα μέτρα, τα μέτρα έγκρισης τύπου για τα οχήματα, του Euro 3, Euro 4 και Euro 5, σε διαβάθμιση, διαδοχικά βήματα. Εδώ ακούσαμε τη γνώμη, όπως κάνουμε και για άλλες κατηγορίες οχημάτων ε, σε ό,τι αφορά την έγκριση τύπου, να έχουμε δηλαδή μια βαθμιαία προσέγγιση. Ο τελικός μας στόχος είναι από το 2020 να έχουμε ε, πιο φιλόδοξες οριακές τιμές για τα οχήματα που να είναι συγκρίσιμες με τα επιβατικά οχήματα. Με τις εκπομπές των επιβατικών οχημάτων. Να πω μάλιστα από τώρα ότι ως αποτέλεσμα της μελέτης αντικτύπου και των διαφόρων ε, άλλων μελετών που κάναμε, θεωρείται ευκταίο ή επιθυμητό το 2016-2017 ε, να κάνουμε μια μελέτη περιβαλλοντική για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ούτως ώστε να ελέγξουμε τα τεχνικά στοιχεία και την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων βημάτων για τον περιορισμό των εκπομπών που θα προκύψουν μέσω της νομοθεσίας, που θα συστήσει η νομοθεσία. Πριν δηλαδή περάσουμε στην ε, τελική φάση των οριακών τιμών, προτείνουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Αυτά τα μέτρα, λόγω της φύσης της έγκριση τύπου, αφορούν τα νέα οχήματα. Και κάτι άλλο που ισχύει και για άλλες κατηγορίες ε, οχημάτων οδικών μεταφορών ε, είναι το θέμα του διοξιδίου του άνθρακα. Σε ό,τι αφορά το διοξείδιο του άνθρακα, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με την πρόταση είναι να δημιουργήσουμε μια πρώτη βάση ούτω ώστε ο νομοθέτης, αν το επιθυμεί, να προβεί στα απαραίτητα νομοθετήματα. Εδώ μιλάμε για την αποτελεσματικότητα, για την εξοικονόμηση μάλλον καυσίμων η εξοικονόμηση των καυσίμων μετριέται τη στιγμή της έγκρισης τύπου και μπορεί να, να συμπεριληφθεί ως ε, ένδειξη. Δεν βάζουμε δηλαδή όριο στο διοξείδιο του άνθρακα, αλλά έχουμε προτείνει κάποιες προϋποθέσεις ενδεικτικά για την κατανάλωση και εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα των οχημάτων. Νομίζω ότι είναι για το καλό των ε, καταναλωτών που με αυτόν τον τρόπο θα λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες και εν πάση περιπτώσει να συγκρίνουν και με άλλα μέσα μεταφορών όταν επιλέγουν τι θα αγοράσουν. Νομίζουμε ότι αυτή είναι μια σημαντική συνεισφορά. για τη βελτίωση για τον εξορθολογισμό των οδικών μεταφορών από περιβαλλοντικής άποψης. Η επόμενη διαφάνεια. Υπήρχαν και άλλε ε, δυνατότητες, άλλε επιλογές ό,τι αφορά τις ε, εκπομπές, τις οποίες εξετάσαμε. ιδίω σε σχέση με τις δοκιμές κύκλου που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση των εκπομπών. Υπάρχουν διά, διάφορες εναλλακτικές λύσεις που μπορούμε να εξετάσουμε, αλλά ως αποτέλεσμα της μελέτης, της μελέτης αντικτύπου υπάρχει μία που συστήνουμε, που συστήνεται μέσω της μελέτης αντικτύπου για την τελική φάση. Είναι η χρήση ενός ενιαίου α, κύκλου δοκιμών για όλα τα οχήματα της κατηγορίας αυτής ΕΛΑ. Είναι θέμα όχι μόνο τεχνικής λογικής, αλλά και απλούστευσης του νομικού πλαισίου σε μια φάση που γίνονται πολλές συζητήσεις για τον κύκλο δοκιμών και για το πόσο ρεαλιστική είναι αυτή. Πιστεύουμε ότι τελικά ε, χρησιμοποιώντας ένα κύκλο δοκιμών που εγκρίνεται και παγκοσμίω. Αυτή τη στιγμή γίνεται δουλειά σε επίπεδο UNESCO με την εμπλοκή όλων των μεγάλων φορέων και ενδιαφερομένων της Ινδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων ακόμη, ούτως ώστε να έχουμε ένα παγκόσμιο τεχνικό κανονισμό για, τις, ε, για τον κύκλο δοκιμών. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν ε, κατά ανάγκη όρια. Κάθε ρυθμιστική αρχή βεβαίως θα επιλέξει, θα καθορίσει, εν όπως θεωρεί, σωστά τα όρια. Αλλά η χρήση ενός ενιαίου τέτοιου κύκλου δοκιμών, όσο πιο ευρέως γίνεται, θα είναι ένα πλεονέκτημα να χρησιμοποιηθεί γενικά, όσο πιο ευρέως. Και τα περιβαλλοντικά μέτρα. Αυτό που θεωρείται σημαντικό είναι η επίδοση του κινητήρα από περιβαλλοντικής άποψης να εξασφαλίσετε μόνο, όχι μόνο τη στιγμή της έγκρισης τύπου, αλλά πιο μακροπρόθεσμα αν γίνεται, για όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, εφόσον είναι εφικτό αυτό. Μεγάλη πρόκληση αυτή. Έχουμε εξετάσει διάφορες επιλογές στη μελέτη αντικτύπου, διάφορες αναλεκτικές λύσεις, για, την καλύτερη, για να δούμε την καλύτερη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ε, διάρκεια και τις προϋποθέσεις διάρκειας και με βάση τη μελέτη αντικτύπου καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η διαβάθμιση αυτών των προϋποθέσεων βάσει στην κατηγορία του προϊόντος είναι η καλύτερη προσέγγιση. Βάσει της κατηγορίας του προϊόντος, λοιπόν. Τώρα μέτρα για την κατασκευή του οχήματος. όσοι συνδέονται και ασχολούνται με τις ε, επιδόσεις εκπομπών γνωρίζουν το, το διαγνωστικό σύστημα που είναι πάνω στον πίνακα ελέγχου. Σημαντικό για, το, για τις εκπομπές αυτό το σύστημα. Και εδώ υπάρχουν διάφορες συναλλακτικές λύσεις που μπορούν να συνδυαστούν. Παραδείγματο χάρη να μην υπάρχει διαγνωστικό σύστημα στον πίνακα ελέγχου, καμία πληροφορία η πρόσβαση στις πληροφορίες ε, διόρθωσης. Δεύτερον, ε, κάποιες ε, διατάξεις που προβλέπονται για τα επιβατικά αυτοκίνητα και η καλύτερη δυνατή τεχνολογία, αυτή που προτείνουμε προτείνουμε να κάνουμε μια πρόταση αναλογική σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, αλλά και το κόστος. Και για την ε, βιομηχανία και για τον κλάδο. Και από την άλλη, να λάβουμε υπόψη μας και την τεχνική πρόοδο που υπάρχει στον τομέα. Πάω τώρα στα συμπεράσματα σιγά σιγά της ε, παρουσίασης. Τα χαρακτηριστικά που καλύπτει ο κανονισμός είναι οι διατάξεις ε, εποπτείας της αγοράς που ανέφερα, η υποχρεωτική χρήση του ABS. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του ABS του προκεχωρημένου ε, συστήματος τροχοπέδης και του ABS, να εγκαταλείψουμε αυτό που προβλέπει ο σημερινός κανονισμός, δηλαδή οι εθνικές αρχές να βάζουν ένα περιορισμό στην ισχύ, ε, περιορισμό ε, στα 74 κιλοβάτ. αυτή, η διάταξη χρησιμοποιείται από τη Γαλλία στο σημερινό κανονισμό και δημιούργησε πολλές αντιδράσεις. Αλλά για να μην μακρηγορώ, νομίζω ότι η μελέτη αντικτύπου και τα δεδομένα που εξετάσαμε καταλήγουν στο ότι η προστιθέμενη αξία ως προς την ασφάλεια δεν συστήνει, δεν να μας σωθούν στο να κρατήσουμε το, αυτή τη διάταξη. Ε, μέτρα κατά του μαστορέματος και ανακατηγοριοποίηση των οχημάτων. Αλλαγή της κατηγορίας. Η σημερινή νομοθεσία θεωρεί ότι όλα αυτά τα οχήματα είναι μία κατηγορία. Τα μίνιο αυτοκίνητα, τα quads, οι τετράτροχες ε, μοτοσυκλέτες και άλλα προϊόντα δηλαδή. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να εξορθολογήσουμε τον κλάδο, να κάνουμε κάποια διαφοροποίηση δηλαδή με σκοπό να αντιμετωπίσουμε πιο στοχοθετημένα τις διατάξει και τις προϋποθέσεις που προτείνουμε για τα προϊόντα αυτά αλλαγή της κατηγορίας, το πέρασμα από μια κατηγορία σε άλλη κάποιων οχημάτων, είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό. Τελευταία διαφάνεια είναι οι συνέπειες της μελέτης αντικτύπου και όλων όσων προανέφερα στην παρουσίασή μου. υποχρεωτική εισαγωγή ενός απλού ε, διαγνωστικού συστήματος στον πίνακα ελέγχου μαζί με προϋποθέσεις για πρόσβαση στην πληροφορία συντήρησης και επιδιόρθωσης, μια βαθμιαία προσέγγιση για την βαθμιαία για να καταστήσουμε ε, βαθμία τις προϋποθέσεις πιο αυστηρές. Ε, ορολογία αντίστοιχη για τα επιβατικά αυτοκίνητα, γύρω 3, γύρω 4, γύρω 5. Στη Γαλλία χρησιμοποιούμε το Euro 4, Euro 5 και Euro 6 για τις μοτοσυκλέτες. Και για όλα τα οχήματα αυτής της κατηγορίας να χρησιμοποιήσουμε ένα κύκλο δοκιμών ε, των ε, εκπομπών Επίσης, ε, υποχρεωτικός φωτισμός. Ανάβουν τα φώτα ε, και τη μέρα, με το που ανάβεται δηλαδή το αυτοκίνητο. Υποχρεωτικό αυτό. Πιστεύουμε ότι αυτόματα το άναμα των φώτων και στα μηχανάκια και στις μοτοσυκλέτες νομίζουμε ότι θα συνεισφέρει στην αύξηση της ασφάλειας αυτών των προϊόντων. Έχω κι άλλα να πω, πολλά να πω, αλλά νομίζω ότι καταχράστηκα του χρόνου σας, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι έτοιμος να απαντήσω και σε όποιες ερωτήσεις έχετε. Ευχαριστώ. Uh, Εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω πως διαθέσαμε μία ώρα και ένα τέταρτο για να κάνουμε μία συγκεκριμένη επισκόπηση μιας πολύ περίπλοκης ε, πρότασης και νομίζω ότι έχουν αρκετά στοιχεία τα λεγόμενά σας τα οποία πρέπει να κατανοήσουμε. Πριν σβήσουν οι διαφάνειες, ε, διαπίστωσα πως το πακέτο που μας έχετε δώσει έχετε και κάποια γραφήματα και θα ήθελα να καταλάβω πόσοι από εμά κατάλαβαν τη διαφορά μεταξύ του συνδυασμένου συστήματος πέδησης και του ABS. Νομίζω πως αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό τεχνικό ζήτημα και επίσης είναι και τελείως διαφορετικό το κόστος των δύο συστημάτων. Δεν ξέρω αν έχετε τις συγκεκριμένες διαφάνειες μαζί. Ε, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε για να εξηγήσετε το θέμα στους συναδέλφους. Πείτε μας λοιπόν αυτά τα συστήματα ακριβώς πώς διαφέρουν μεταξύ τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Περάστε λοιπόν στη διαφάνεια 21. Με συγχωρείτε, 29 διορθώνει ο μιλητής. Κοιτάξτε τη διαφάνεια 29. Έχετε εδώ λοιπόν ένα σχεδιάγραμμα με τα διάφορα συστήματα πέδησης που υπάρχουν. Αριστερά λοιπόν έχετε το συμβατικό σύστημα όπου για τις ε, μηχανές για παράδειγμα έχετε ένα μοχλό ε, που καλύπτει το μπροστινό φρένο και ένα πετάλι στα χέρια στις ε, λαβίδες αυτό και ένα ε, πετάλι που, καλύγει, ε, που καλύπτει τα δύο κυκλώματα πίσω και χρησιμοποιούνται ξεχωριστά τα δύο αυτά, το εμπρόσιο και το πίσιο φρένο. Αυτή είναι η τεχνολογία και μπορείτε αυτά να τα συνδυάσετε με διάφορα επίπεδα διαφορετικά μεταξύ τους έτσι ώστε να έχετε για παράδειγμα ένα σύστημα που ενεργοποιείται ένα πραγματικό φρένο, το πίσω, το πίσω φρένο ε, και παράλληλα να φρενάρεται και τον ε, ευρωστιό ε, τροχό. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα κύκλωμα όπου χρησιμοποιεί κανείς το πετάλι για να φρενάρει πίσω και παράλληλα με τον τρόπο αυτό ενεργοποιεί και τον μπροστινό τροχό. Ένα ακόμα προθυμένο στοιχείο και μιλάμε πάντα για τη συνδυασμένη υπέδηση είναι είτε να χρησιμοποιήσει κανείς κάποιο από τα δύο που έχει στη διάθεσή του Δηλαδή είτε με το πετάλι είτε με το σύστημα στα χέρια να μπορεί να μπροκάρει τον πίσω ή τον προστινό τροχό. Ίσως αυτό δεν φαίνεται από τα σχέδια που σας έχουμε δώσει. Αυτό λοιπόν είναι το συνδυασμένο σύστημα. Χρησιμοποιώντας λοιπόν ένα από τα δύο ε, εργαλεία που προσφέρονται, είτε δηλαδή το μοχλό που έχετε στο τιμόνι, είτε το πετάλι που έχετε χαμηλά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ε, και τον μπροστινό φρένο και το φρένο στον πίσω τροχό. Περνάμε λοιπόν ε, στο σύστημα που είναι το γνωστό ABS, όπου δεν έχουμε κλείδωμα των τροχών. Μιλάμε εδώ για μια ηλεκτρονική εντολή που ενεργοποιεί και αυτό βέβαια βασίζεται σε μια σειρά παραμέτρους, ενεργοποιεί και το εμπρόστιο και το πίστιο φρένο. Ε, ο ίδιος ο υπολογιστής ε, αποφασίζει σε ποιο βαθμό τα μπλοκάρει και δίνει μια προστιθέμενη αξία σε σχέση με το συνδυασμένο σύστημα πέδησης γιατί έχει αυτή την ε, λειτουργία anti-lock, δηλαδή δεν κλειδώνουν οι τροχοί. Το σύστημα λειτουργεί με έναν τρόπο που είναι γνωστός ήδη από τα αυτοκίνητα. Αν λοιπόν είτε ο μπροστινός τροχός είτε ο πίσω τροχός κλειδώνει, ε, το σύστημα μετριάζει την πίεση που οδηγός, ε, με την οποία ο οδηγός πατάει το φρένο έτσι ώστε οι τροχοί να μην κλειδώσουν. Αυτή είναι η βασική διαφορά με το συνδυασμένο σύστημα και αν περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι δεν έχω να σας πω κάτι παραπάνω. Η βασική ιδέα την οποία έχουμε αναλύσει εδώ στην μελέτη αντικτύπου είναι κατά πόσο χρειάζεται τέτοιου είδους συστήματα δηλαδή προηγμένης τεχνολογίας να χρησιμοποιούνται και αν ναι, σε ποιο βαθμό και μάλιστα για ποια κατηγορία προϊόντων θα χρειάζονταν κάτι τέτοιο που θα ήταν λογικό. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε ήταν πως η προσέγγιση που θεωρούμε να είναι η πιο ενδεδειγμένη είναι αυτή την οποία προτείνουμε βέβαια και στο κείμενο που έχουμε υποβάλει. Νομίζω πως το θέμα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για όλους και είμαι σίγουρος πως οι βουλευτές θα υποβάλουν σχετικές ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βάντερ Κάμπ έχει να κάνει μια παρουσίαση. Κάντε την παρουσίασή σας και μετά θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις και για τις δύο παρουσιάσεις. Συμφωνείτε, βεβαίως. Ωραία, λοιπόν. Εδώ θα δούμε ε, το απόγευμα και άλλες διαφάνειες. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που σας δίνω το λόγο. Και αφού τελειώσετε κι εσείς, ε, ερωτήσεις είτε προς την Κομισιόν είτε προς τη δική σας παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω ποιος θα ενεργοποιήσει ε, τις διαφάνειες για να τις δούμε μία-μία και με τη σωστή σειρά. Κύριε Πρόεδρε, δεν ήμουν σίγουρος κατά πόσο θα ήταν φυσιολογικό ο εισηγητής να κάνει μία ε, μακροσκελή παρουσίαση και Εάν δεν συνηθίζετε κάτι τέτοιο, είμαι εγώ ο πρώτος που θα πάρει το λόγο για ώρα σήμερα το απόγευμα. Να, μια καινοτομία που μπορώ να σας προσφέρω. Να σας πω πάντω πως με την ιδιότητα του εισηγητή στηρίζω, στηρίζω την βούληση αυτή βελτίωση και απλούστευσης του νομοθετικού πλαισίου. Ε, νομίζω πως μας προετοιμάζουν για τα Χριστούγεννα. Έτσι είναι πραγματικά ζεστή ατμόσφαιρα με αυτό το φωτισμό, λέει ο μιλητής. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και την κυρία Ρούλ γιατί αυτό που επιθυμούμε εμείς είναι να μειώσουμε τις εκπομπές, τις εκπομπές αερίων που ρηπαίνουν. Και για τα δίτροχα να σας πω πως οι εκπομπές τους είναι τεράστιες. Μπα, πέρασαν τα Χριστούγεννα, λέει ο μιλητής. Ανάψανε και πάλι τα φώτα. Μπορείτε να τα ξανασβήσετε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, περνάμε στην τρίτη γραμμή που είναι η διάσταση της ασφάλειας η οποία επίσης για μας είναι σημαντική. Τουλάχιστον αυτό μας εξήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε λοιπόν 5.200 θανάτους ετησίους. Νομίζω πως ο αριθμός αυτός είναι τρομακτικός. Και τι σημαίνει όταν έχουμε αεροπορικό δυστύχημα, ο αριθμός θανάτων είναι πολύ πιο περιορισμένος. Αυτά σας τα λέω για να κάνετε μια σύγκριση. Θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε ένα καλύτερο επιμερισμό αυτών των στοιχείων, γιατί έχουμε βέβαια συλλέξει όλα τα τροχέα από την Δανία μέχρι τη Σαρδινία και νομίζω πως τα στοιχεία αυτά καταρχήν ε, είναι εντυπωσιακά, θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε μια κατανομή για να δούμε σε τι ακριβώς αντιστοιχούν αναχώρα, ανα είδος ατυχήματος. Ε, στον κανονισμό που ετοιμάζουμε θα πρέπει να δοθούν κάποιες νέες ευκαιρίες χρησιμοποιώντας με καλύτερο τρόπο την τεχνολογική πρόοδο και την τεχνολογική καινοτομία. Και θα επανέλθω βέβαια στη σημασία την οικονομική σημασία που έχει ο, ο κλάδος των δίτροχων στην Ευρώπη. 30 δις εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, με συγχωρείτε 34 δις το χρόνο, 159.000 απασχολούμενοι και 25 από αυτούς στον κατασκευαστικό κλάδο. Και για τα 4x4 ε, έχουμε ή 12.000 ε, απασχολούμενους και για τα ΜΙΚΑΡ 340.000 οχήματα με 20.000 εργαζόμενους στον ε, κλάδο. Η επόμενη διαφάνεια. Θα διαπιστώσετε πως έχουμε πάνω από 800 επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό, δηλαδή κατασκευάζουν δίτροχα οχήματα, με κύκλο εργασιών 8 εκατομμυρίων ευρώ συνήθως. Το 80% είναι εγκατεστημένες σε έξι κράτη-μέλη, στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Αυστρία. Ποια είναι λοιπόν τα σημεία τα οποία χρειάζεται εμείς να συζητήσουμε, γιατί νομίζω ότι θα γίνει όντως συζήτηση σήμερα το απόγευμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στοχεύει στο να εφαρμόσει από την 1η Ιανουαρίου του 2013 τον κανονισμό. Κατά τη γνώμη μας αυτό είναι υπερβολικά φιλόδοξο θα μπορούσε να μας δώσει και κάποιες προφορίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί, γιατί υπάρχει μία σειρά ρυθμιστικών βημάτων που θα πρέπει να ακολουθηθεί το 2012 έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για το 2013. Να ρωτιέμαι λοιπόν, αν πραγματικά θα προλάβουμε και για τον λόγο αυτό θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή όλων εδώ και αναφέρομαι και στους κοιόδης εισηγητές, αν υπάρχει σχέση και σύνδεση μεταξύ αυτού του κανονισμού και άλλων οδηγιών ή κανονισμών ε, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα σκαριά και έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια και πιο συγκεκριμένα με την επιθεώρηση και την έγκριση τύπου οχημάτων γιατί όλα αυτά σχετίζονται με άλλες, όπως σας είπα και προηγουμένως, οδηγίες. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν, εμείς ως νομοθέτες στο πληθυντικό, να δούμε πώς συνδέονται μεταξύ τους οι διάφοροι κανονισμοί που ήδη είναι σε ισχύ. Με την ιδιότητα του εισηγητή έχω την πρόθεση να κάνω και μια σειρά επισκέψεων ε, ε, επιτόπου με τους ε, σκιώδεις εισηγητές και ελπίζω πως οι συνάδελφοι θα καταφέρουν να έρθουν και θα απελευθερωθούν από τα καθήκοντά τους. Στις 28 Ιανουαρίου θα πάμε στο Λέλισταντ των κάτω χωρών και επίσης θα επισκεφθούμε την Έση δίπλα στο Ρήνο. Και μετά 23 με 25 Φεβρουαρίου θα πάμε σε, τρεις, ε, σε τρία εργοστάσια στην Ιταλία και θα επισκεφτούμε και μία επιχείρηση Ιαπωνικών συμφερόντων εκεί. Αυτό λοιπόν είναι το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθήσουμε. Έχουμε λοιπόν καταρχήν τις ε, επισκέψεις. Είναι πολύ σφιχτές οι προθεσμίες, αλλά είμαι πάντα αισιόδοξο και φιλόδοξο και νομίζω πως δεν θα πρέπει αυτό το νομοθετικό έργο να καθυστερήσει. Θα κάνω λοιπόν ό,τι μπορώ με τους χειώδες εισηγητές για να σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα αυτό που επαναλαμβάνω είναι εξαιρετικά απαιτητικό. Μπέρναμε στην επόμενη διαφάνεια. Α, δεν έχουμε άλλη. Κύριε Πρόεδρε, ως συμπέρασμα λοιπόν, και σας παρακαλώ να ανάψετε και πάλι τα φώτα στην αίθουσα, ο πρόεδρος θα σας διακόψω, αλλά για όσους μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο, δεν μπορούσαν να δουν τις διαφάνειες ε, σκοτάδι. Το μόνο που έβλεπαν ήταν το κόκκινο φως από το μικρόφωνο σας. Για όποιον λοιπόν μας παρακολουθεί μέσω διαδικτύου, στείλτε μας ένα email για να σας στείλουμε εμείς τις διαφάνειες αν ενδιαφέρεστε. Ωραία, λοιπόν, ανάψανε και πάλι τα φώτα να απευθύνω και κάποιες ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Λοιπόν, για το θέμα αυτό και για την παρουσίαση που έγινε, πρέπει να σε εξομολογηθώ πως υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία δεν τα κατάλαβα. Ποιες είναι οι κατηγορίες οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής για τις ε, μηχανές με τέσσερις ρόδες, τις αποκαλούμενες γουρούνες, ε, έχω να ρωτήσω το εξής στην Κομισιόν. θεωρείται πως δεν ανήκουν. Αντίθετα, θεωρείται πως εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Νομίζω ότι για την ευρωπαϊκή κοινωνία αυτό αποτελεί μια τεράστια πρόκληση. Μιλάμε για, το, ε, για αυτή την καινοτομία, το, το ηλεκτρικό ποδήλατο και θα ήθελα να μου πείτε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί το έχετε συμπεριλάβει στο κείμενο ενώ ε, οι τετράτροχες μηχανές δεν έχουν συμπεριληφθεί. Και θα ήθελα να μου δώσετε και κάποιες πληροφορίες για το κόστος του συστήματος ABS. Ε. Ξέρω βέβαια πως το κόστος είναι μεγάλο για τις εταιρείες, αλλά λόγω μαζικής παραγωγής φαντάζομαι πως το... η τιμή θα πρέπει να πέσει. Ε, αυτές τις ερωτήσεις είχα και θα ήθελα να τις απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Όσον αφορά τώρα τα αυτοκίνητα εκτός αυτού του ε, πλαισίου, ε, είδαμε τις διαβάνεις και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό απαντώνται τα ερωτήματα, αλλά ίσως μπορείτε κι εσείς να τοποθετηθείτε σε ορισμένες από αυτές. Θα ήθελα να φερθώ κυρίως ε, στα οχήματα που έχουν ως στόχο που έχουν κατασκευαστεί για να ε, ε, λειτουργούν, να ε, τρέχουν εκτός δρόμου. Τα off-road όπως λέμε. Έχουμε εδώ αρκετούς ε, σκιώδεις αλλά νομίζω ότι δεν είναι κανείς εδώ από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Κυρία Ρούλα είναι εδώ. Ε, θα ήθελα να δώσω λοιπόν το λόγο και ίσως μπορεί να τοποθετηθεί και μετά η κυρία Κόπολα. κυρία Ρούλα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και βεβαίως και την ε, Κομισιόν για τις ε, πληροφορίες που μας έδωσαν και ήταν πραγματικά μια πολύ καλή εισαγωγή. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η εισαγωγή πράγματι θα ήταν πολύ δύσκολο να μπορέσει κανείς να αποκτήσει μια εικόνα σε αυτό το τόσο τεχνικό θέμα. Και εγώ θέλω να κάνω περίπου μια ερώτηση που κάνατε κι εσείς. Ρωτήσαμε ποιοι τύποι περιλαμβάνονται, ποιοι όχι και γιατί. Η απάντηση δεν είναι απόλυτα σαφής. Διαβάζω λοιπόν τι εξηγήσει που μα εδόθησαν. σω μπορείτε εσεί να μα το εξηγήσετε βέβαια προφορικά γιατί ορισμένοι τύποι αυτοκινήτων δεν περιλήφθησαν και ποιοι περιλήφθησαν. Γιατί όταν γίνεται μία απλούστευση είναι πολύ δύσκολο να υπάρχουν εξαιρέσει. γιατί αυτό περιπλέκει ακόμα ε, το θέμα περαιτέρω. Αυτή ήταν η βασική μου ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, η πρώτη μου ερώτηση είναι ρητορικής φύσεως. Υπάρχουν εδώ άνθρωποι σε αυτή την αίθουσα που να οδηγούν μοτοσυκλέτα. Μήπως υπάρχουν και από τους ρυθμιστές, από όσου κάνουν την νομοθεσία, άνθρωποι που να οδηγούν επίσης νομοσυκλέτα για να ξέρουν ποια είναι τα θέματα κλειδί. Ένα θέμα κλειδί είναι κατά πόσον τα μέτρα αυτά θα έχουν οποιαδήποτε σχέση με μεγαλύτερη ασφάλεια. Θα οδηγήσουν, εν σε μεγαλύτερη ασφάλεια. Και από ό,τι κατάλαβα, άκουσα ότι οι ίδιοι μοτοσυκλετιστές ανησυχούν ε, όσον αφορά σε αυτή την πρόταση. Γιατί συνεπάγεται μεγάλες δαπάνες, αλλά δεν οδηγεί σε μεγαλύτερη ασφάλεια. Άρα δηλαδή πρόκειται για λάθος επένδυση. Αν δεν την προσαρμόσουμε λιγάκι, θα ισχύσει αυτό που σας είπα. Θα αναφέρω και ένα παράδειγμα. Το υποχρεωτικό σύστημα αναφέρθηκε το υποχρεωτικό σύστημα EBS και το διαγνωστικό σύστημα που θα πρέπει να υπάρχει στον πίνακα ε, στον πίνακα ελέγχου. Διερωτώ με τι είδου συνέπειε θα υπάρχουν. Θα υπάρχουν νέα όρια εκπομπών, ε, νέε απαιτήσει ε, για ε, τη βενζίνη, για το τάγκ τη βενζίνη. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Θα σημαίνουν άραγε και νέους περιορισμούς σχετικά με το μετριασμό και τις τροποποίησεις. Και όσον αφορά τις συνέπειες. Ε, μήπως θα αυξηθούν και οι τιμές των μοτοσυκλετών λόγω των νέων αυτών ε, προδιαγραφών. Τέσσερα δις ανά δέκα χρόνια. Και αυτό σημαίνει μονοπόλιο. Το κόστος αυτό ε, κατ' ουσίαν είναι πολύ μεγάλο για τις μικρές εταιρείες και οδηγεί σε μονοπόλια. Με ανησυχεί λιγάκι το θέμα της προσαρμογής. Εμένα, εγώ αγαπώ τους άντρες και νομίζω ότι σε κάθε άντρα κρύβεται και ένας μηχανικός που του αρέσει να πειράζει εισαγωγικά και να τροποποιεί το αυτοκίνητό του. Να μαστορεύει πάνω σε αυτό. Εσείς ε, πιστεύετε ότι αυτό το πείραγμα εισαγωγικά είναι επικίνδυνο, πείραγμα της μηχανής. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη αξιολόγηση των συνεπειών και αν γίνει βέβαια κάτι τέτοιο, πάρα πολλοί άντρε τελικά ε, δεν θα μπορούν να έχουν χόμπι. Φαντάστε λοιπόν τι τραγική η κατάσταση αυτή για του άντρε. Και γιατί να τους ε, αφαιρέσουμε αυτό το χόμπι αν ε, δεν επιτύχουμε τίποτα, καμία βελτίωση. αυτή είναι η ανησυχία μου και αυτό ήθελα να πω. Thank you, Um, Heidi. Κοιτάξτε, το θέμα τη ασφάλεια αυτό ίσω μπορεί να το αιτιολογήσει η Κομισιόν. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν ξεκάθαρα ότι ε, τα ε, ατυχήματα με μοτοσυκλέτες είναι τα πλέον θανατηφόρα που λαμβάνουν χώρα και αυτά αφορούν κυρίως νέους άνδρες. Γι' αυτό λοιπόν διαρωτώ με. Ε, αν πρόκειται να, να προκύψει βελτίωση, θα το έβρισκα καλό. Δεν πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε χόμπι να είναι και θανατηφόρα. Και από την άλλη, όπω ε, προτείνει η Κομισιόν, ε, θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι ενιαίες οι προδιαγραφέ σε ολόκληρο τον κόσμο γιατί όταν πήγαμε στην Ινδία είδαμε ότι οι Ινδοί χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τη μοτοσυκλέτα και αυτό έχει πολύ μεγάλες συνέπειες στο περιβάλλον. Εκεί λοιπόν το θέμα των εκπομπών είναι τραγικό και ως εκ τούτου αν είχαμε ενιαίες παγκόσμιες προδιαγραφές σε όλο τον κόσμο αυτό θα ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Λοιπόν, τώρα θα σας μιλήσω ως ε, σκιώδης ηγητής της πολιτικής ομάδας και θα ήθελα να επαναφέρω ορισμένα θέματα που είπα και σήμερα το πρωί για να υπάρχει έτσι κάποια συνέπεια. Το πρώτο έχει σχέση με τα ανταλλακτικά. Όταν λοιπόν δουλέψαμε πάνω στην οδηγία για τα οχήματα, για τα αυτοκίνητα, αυτό είναι ένα θέμα που προκαλεί τη σύγχυση. Και οι εταιρείε κατ' ουσίαν ικανοποιήθηκαν που έχουν ένα νέο πλαίσιο για την έγκριση τύπου και ήταν απόλυτα έτοιμες να ε, δοκιμαστούν τα προϊόντα τους, ε, τα ανταλλακτικά, ε, για να μην επιδεινωθεί το θέμα της ασφάλειας των αυτοκινήτων. Επίσης, ε, οι κατασκευαστές ε, των αυτοκινήτων ε, δυστυχώς διαπίστωσαν ότι δεν μπορούν να πουλήσουν αυτά τα ανταλλακτικά και έτσι λοιπόν προέκυψε μια πολύ μεγαλύτερη αγορά από ό,τι υπήρχε κατά το παρελθόν. Νομίζω λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να επιτρέψουμε να λάβουν χώρα τέτοιου είδου διαδικασίες. Δεύτερον, όσον αφορά στο θέμα της διαθεσιμότητας των τεχνικών πληροφοριών. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί εδώ μιλάμε, κυρίως όταν μιλάμε για ακριβά αυτοκίνητα, ε, τα οποία ε, επισκευάζονται σε μικρά συνεργεία. Εκεί το θέμα της διαθεσιμότητας των πληροφοριών είναι καθοριστική σημασίας. Εάν αυτά τα δεδομένα υπάρχουν σε ευκολόχρηστη μορφή, τότε και οι άνθρωποι δεν θα είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσουν ακριβά λογισμικά. Αυτά όσον αφορά στις εκπομπές. Και κάτι άλλο που θέλω να πω έχει σχέση με τα ε, με το με τις μοτοσυκλέτες. Χάρηκα πάρα πολύ που η μελέτη αντικτύπου της ε, Κομισιόν δεν αναφέρει περιορισμό ε, της υποδύναμης των μοτοσυκλετιστών των Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν οπωσδήποτε να περιστεί αυτή η υποδύναμη. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι σημαντικό και αυτό είναι κάτι ε, ε, για το οποίο μπορούμε να καθησυχάσουμε τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα μοτοσυκλέτες ότι πράγματι ελήφθη υπόψη. Ας πάμε στο θέμα της ασφάλειας. Εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον θέμα που το θίξατε δηλαδή ποιες ε, κατηγορίες μοτοσυκλετών έχουν ε, σύστημα ABS και ποιες έχουν σύστημα αντιεμπλοκής, προηγμένο σύστημα αντιεμπλοκής και τι γίνεται με τις δαπάνες ή ε, τι γίνεται με τα στατιστικά δεδομένα. Νομίζω ότι το ευρύτερο θέμα, ίσως επ' αυτού μπορείτε λιγάκι να τοποθετηθείτε, αφορά στα θανατηφόρα ατυχήματα με μοτοσυκλέτες. Δεν ξέρω αν με παρακολουθείτε, γιατί αυτό που λέω έχει σχέση με αυτά που είπατε κι εσείς. Λοιπόν, όσον αφορά στο θέμα ε, θανατηφόρων ατυχημάτων, ποια είναι η σχέση ανάμεσα στο να χάσει κανείς τον έλεγχο στην, ε, κατά το φρενάρισμα, κατά την πέδηση και το μοιραίο της υπόθεσης γιατί αυτό έχει σχέση με την απόφαση που πρέπει να ληφθεί σχετικά με τα δεδομένα. Σε αυτόν το συγκεκριμένο τομέα, ε, νομίζω είμαστε πεπισμένοι ότι όσον αφορά την βελτίωση τη ασφάλεια, υπάρχει σαφή συσχετισμό μεταξύ αυτών των δύο στοιχείων. Και νομίζω ότι αυτό είναι και πιθανό, γιατί αν είναι μπροστά το σύστημα φρεναρίσματος, ο μοτοσυκλετιστής πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερες ικανότητες από την περίπτωση που έχει σύστημα φρεναρίσματος μπρος και πίσω. Και εγώ δεν οδηγώ μοτοσυκλέτα ο ίδιος, αλλά αντιμετωπίζω αυτό το θέμα με τα αυτοκίνητα. Επειδή λοιπόν πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα όσον αφορά ε, το κόστος ανάπτυξης, το κόστος ε, των μοτοσυκλετών ε, και της πρόσβασης στα δεδομένα, θα ήταν χρήσιμο να μας πείτε περισσότερα πράγματα, γιατί είδα λιγάκι τη μελέτη αντικτύπου για να βρω αυτά τα στοιχεία τα στοιχεία που μας παρουσιάζονται είναι σαφώς εύληπτα, αλλά δεν βρίσκω την απάντηση που θέλω. Και το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Έχει σχέση και πάλι με την ασφάλεια. Νομίζω ότι, κατά την άποψή μου, υπήρξαν πολλές ε, ε, ανησυχίες για την ασφάλεια των πολύ ελαφρών οχημάτων. Και ε, δημοσιεύτηκαν crash test πάρα πολλά για αυτά τα ε, ελαφρά αυτοκίνητα και τα αποτελέσματα ήταν πολύ δυσάρεστα. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες σχετικά ε, με ατυχήματα που έγιναν με αυτά τα ε, ελαφρά οχήματα. Μήπως μπορείτε λιγάκι να μας το εξηγήσετε, γιατί ο τρόπος κατασκευής αυτών των μικρών οχημάτων είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν με τον οποίο κατασκευάζονται οι μοτοσυκλέτες. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, όσον αφορά στο θέμα της ασφάλειας, αυτά τα ελαφρά και πολύ ελαφρά οχήματα, τι σημαίνει, τι γίνεται στην ασφάλεια σε αυτά τα οχήματα σε σχέση με τις μοτοσυκλέτες. Ίσως μπορείτε να μας το απαντήσετε. Mrs. Anybody got any other questions in the first round for the Commission? Okay, so can I invite you to respond to the first round of questions? And if we have time, certainly I'll give Mr. Van der Kamp the opportunity to sum up. But um, let's hear. Λοιπόν, ας ακούσουμε από την Επιτροπή καταρχήν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και όσους υπέβαλαν τις ερωτήσεις τους. Θα ήθελα να απαντήσω σε ερωτήσεις ε, σχεδόν με τη σειρά που παρουσιάστηκαν και βεβαίως υπάρχει ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι έθιξαν αρκετά μέλη είναι το θέμα του πεδίου. Αν είναι τεχνικά εφικτό να με βοηθήσετε με τις διαφάνειες θα έλεγα να κατεβάσετε τη διαφάνεια υπαριθμών 20, η οποία ανακεφαλαιώνει όσα δεν αναφέρονται ε, στο πεδίο της ε, πρότασης. Αυτό που δεν αναφέρεται στο πεδίο της πρότασης είναι κατά κύριο λόγο τα οχήματα τα οποία προβλέπονται αποκλειστικά και μόνο για κανονικούς δρόμους, τα άλλα που είναι για off-road, on-road ε, αγώνες, τα αγροτικά αυτοκίνητα, γιατί αυτά καλύπτονται από άλλη πρόταση, αλλά ίσως πρέπει να σκεφτούμε και ε, κάποια άλλα θέματα που αφοράν στα ε, αυτοκίματα παντός εδάφους. Υπάρχουν ε, οι αποκαλούμενες συσκευές αυτορυθμιζόμενες και εδώ το πιο συνηθισμένο προϊόν είναι το Segway. Ίσως το γνωρίζετε μερικοί από εσά. Τα αυτοκίνητα, τα οχήματα, ε, τα οποία και αυτά δεν ε, έχουν τουλάχιστον ένα κάθισμα, αυτά, εν πάση περιπτώσει, είναι τα οχήματα τα οποία αποκλείονται, ρυθμίζονται αλλού. Και νομίζω ότι σα εξήγησα και τι ακριβώ περιλαμβάνεται στο πεδίο τη οδηγία. Μία από τι ερωτήσει που ετέθησαν ε, νομίζω ότι είχε σχέση με του ηλεκτρικού κύκλου. Αυτό που εμεί ε, περιλαμβάνουμε είναι κύκλοι ισχύω, οι οποίοι φτάνουν μέχρι το 1 κιλοβάτ και μέχρι 25 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτό το κάνουμε γιατί αν δούμε λιγάκι τα στοιχεία διαπιστώνουμε ότι η εμφάνισή του στην αγορά, η εμφάνιση αυτών των αυτοκινήτων στην αγορά ήταν πολύ επιτυχημένη, τεράστια η επέκτασή τους. Ε, αυτά λοιπόν, ε, άμα ποδήλατα, αυτά τα ποδήλατα διεδόθηκαν με πολύ μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και τα περίφημα τα είδος pedestrians, Εκεί παρουσιάζεται μια διαφορά στην ταχύτητα, αλλά η διαφορά είναι τέτοια η οποία ε, μεταξύ άλλων μπορεί να αποτελεί και απειλή για την ασφάλεια. Αυτός λοιπόν ο βασικός λόγος γιατί στην ε, κείμενη νομοθεσία δεν περιλάβαμε κύκλους ισχύω μέχρι κάποιο ε, όριο, ανώτατο όριο. Η άλλη ερώτηση αφορούσε τα ε, οχήματα παντός εδάφους. Εδώ κατ' ουσίαν μιλάμε για την ίδια κατηγορία όπως τα τετράτροχα και άλλα αυτοκίνητα. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια ε, ιδιομορφία. Αυτές οι μοτοσικλέτες σε πολλές ε, χώρες ε, χρησιμοποιούνται ως ε, μοτοσικλέτες. Τα τετράτοχα χρησιμοποιούνται ως μοτοσικλέτες με τη μορφή αυτή και σε αστικές περιοχές. Εδώ λοιπόν πλουστεύω λιγάκι την κατάσταση, αλλά χρησιμοποιούνται κυρίως ως ε, οχήματα on roads για αναψυχή. Και κατ' ουσίαν εδώ αντιμετωπίζεται η ίδια πρόκληση όσον αφορά ε, την ασφάλεια, της εκπομπές όπως και στις μοτοσικλέτες. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι κάποια από αυτά τα τετράτροχα οχήματα all terrain όπως λέγονται χρησιμοποιούνται καθαρά και μόνο για γεωργική χρήση off-road σε ανώμαλους δρόμους. Ίσως λοιπόν μπορούμε ε, να ε, σκεφτούμε το θέμα της ε, νομοθεσίας αν βρούμε κάποια λύση για τα γεωργικά οχήματα, ίσως μπορούμε να ρυθμίσουμε και αυτά τα οχήματα ATV που χρησιμοποιούνται σε ανώμαλους δρόμους, off-road, και που δεν καλύπτονται από αυτήν την οδηγία. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το εξής. Ε, κατ' ουσίαν εδώ μιλάμε για αυτά ε, τα τετράτροχα παντός εδάφους. Και εκεί υπάρχουν βέβαια κάποιες σκέψεις όσον αφορά τη σχέση κόστους κόστους-οφέλους. Ε, πράγματι υπάρχει προσθέμενη αξία, ε, θα προκύψει για τους κατασκευαστές κάποια, κάποιο όφελος εάν έχουν έγκριση τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι εθνική έγκριση τύπου. Το άλλο θέμα που ετέθη σε αρκετές ερωτήσεις έχει σχέση με την πρόταση σχετικά με το ABS και το anti-lock ε, το σύστημα ABS και το σύστημα anti-lock και ε, κατ' ουσία προτρέχω γιατί θα μπορούσε να τεθεί ένα ερώτημα σχετικά ε, πού πρέπει να τοποθετηθεί το όριο. Καταρχήν, όσον αφορά το κόστος, εδώ προκύπτουν διάφορες διαπάνε. Κάναμε μία ανάλυση για το ίδιο το ε, σύστημα ABS και πρέπει να σας πω ότι μέσα σε αυτό το σύστημα, στο ABS, και εδώ μιλάω για συστήματα αντιεμπλοκή, αν θέλετε, anti-lock, που έχουν διάφορα χαρακτηριστικά αυτά τα συστήματα. Άρα δηλαδή έχουμε μία βεντάλια, ένα φάσμα πολύ μεγάλο από 50 μέχρι εκατοντάδες ευρώ που μπορεί να κοστίσει το σύστημα αυτό. Βεβαίως δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το κόστος που προστίθεται σε επίπεδο κατασκευαστών αυτό το κόστος για τους κατασκευαστές για να προσαρμόσουν τα υπάρχοντα μοντέλα ή νέες μοτοσικλέτες να εξοπλιστούν και αυτές με αυτό το σύστημα. Πιστεύω λοιπόν ότι το σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε εδώ υπόψη μας αντί για το κόστος του ίδιου του συστήματος είναι ο λόγος. Και αν δούμε το όφελος από την εφαρμογή των μέτρων και τη μελέτη αντικτύπου διεπιστώνουμε ότι υπάρχει ένας λόγος κόστους κόστους-οφέλους της τάξης του 1 προς 3. Έτσι λοιπόν το όφελος αν θέλετε είναι τριπλάσιο σε σχέση με το κόστος και ω εκ τούτου με και αυτή τη ευκαιρία για να απαντήσω και σε μια άλλη ερώτηση. Πράγματι είμαστε ακράδαντα πεπισμένοι ότι παρά το επιπρόσθετο οριακό κόστος το όφελος από τα χαρακτηριστικά αυτού του συστήματος όσον αφορά στην ασφάλεια είναι πολύ μεγάλο. Γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας Μάλλον, να το πω αλλιώς, ε, πράγματι ε, εξετάσαμε πάρα πολλές μελέτες για ατυχήματα και κυρίως ατυχήματα που αφορούν σε δίτροχα. Ο ανθρώπινος παράγων είναι καθοριστική σημασία στην περίπτωση ατυχήματος και ο ανθρώπινος παράγων είναι εκείνος που καθορίζει την περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Εύχομαι κανείς από εμά, αλλά μας ίσως κάποιοι να αντιμετωπίσουν τέτοια έκτακτη ανάγκη. Σε τέτοια περίπτωση πατάει κανείς πολύ απότομα το φρένο που σημαίνει ότι χάνει κανείς τον έλεγχο για διάφορους λόγους. Χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αυτό ισχύει για τα αυτοκίνητα, πόσο μάλλον για τις μοτοσυκλέτες. Ε, υπολογίστηκε λοιπόν ότι μπορούν να σωθούν 6.000 ζωές σε διάρκεια 10 ετών με τη χρήση αυτού του συστήματος. Αν σκεφτούμε πιο συγκεκριμένα τις πόλεις, ακόμα και οι τραυματισμοί κοστίζουν πάρα πολύ στην κοινωνία. Πέρα από το τι υφίσταται ο ίδιος ε, ο άνθρωπος που τραυματίζεται. Το τι σημαίνει για την κοινωνία αυτό οπωσδήποτε πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου σας, αλλά θα ήθελα να περάσω σε κάποια άλλα θέματα που ετέθησαν. Το ένα αφορά στα ανταλλακτικά, όπου εκεί πράγματι θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι όσον αφορά την προσέγγιση για τα ανταλλακτικά. Η δική μας η προσέγγιση είναι συνεπής με αυτά που έχουμε προτείνει σε άλλες ε, νομοθετικές διατάξεις ε, έγκρισης ε, τύπου. Ακούσαμε σήμερα το πρωί για τα αγροτικά. Τώρα, όσον αφορά το όριο των εκπομπών Κοιτάξτε, νομίζω ότι το να επιτύχουμε ε, κάποιο ανώτατο όριο, αυτό είναι ε, πολύ φιλόδοξο, αλλά τελικά αν αρχίσουμε να διαπραγματευόμεθα σε παγκόσμιο επίπεδο, αν λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές του κόσμου που δεν είναι τόσο ε, προηγμένες ως εμείς, αν επιδιώξουμε κάτι τέτοιο, αυτό θα σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κατέβει πάρα πολύ να ε, προτείνει συμβασμούς που για να μας ειλικρινείς δεν είμαστε αυτή τη στιγμή έτοιμοι να τους δεχτούμε. Αυτά όσον αφορά τις ε, εκπομπές ε, και τις οδικές μεταφορές. Τώρα, πάμε στο θέμα, γιατί ετέθη επίσης ένα θέμα σε σχέση με την μετατροπή των αυτοκινήτων, την προσαρμογή τους Νομίζω αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, είτε μας αρέσει είτε όχι, εδώ έχουμε να κάνουμε πολύ περίπλοκα προϊόντα. Προϊόντα όπου ο ηλεκτρονικός έλεγχος ε, παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο. Γι' αυτό λοιπόν το να πειράξει όπως λέμε κανείς τα ηλεκτρονικά στοιχεία, το ηλεκτρονικό πίνικα ενός οχήματος, αυτό συνεπάγεται σοβαρότατους κινδύνους τόσο για την ασφάλεια του οδηγού όσο και για τις εκπομπές. Μπορεί να είναι απόλαυση, αλλά με συγχωρείτε, η πρώτη απόλαυση πάνω απ' όλα είναι να οδηγεί κανείς τη μοτοσικλέτα. Και εδώ ε, θέλω να σας πω, να σας καθησυχάσω, ότι όχι μόνο είμαστε σε ε, συνεργασία, στενή συνεργασία με τους ε, μοτοσικλετιστές, αλλά και στην υπηρεσία μας και εγώ είμαι οδηγός μοτοσικλέτας Άρα δηλαδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτά τα θέματα, το πείραγμα ή το μη πείραγμα είναι καθοριστική σημασίας εφόσον επιθυμούμε να διασφαλίσουμε όλα τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου ή του οχήματος με συγχωρείτε κυρίως σε μοτοσυκλέτες αναφέρομαι όπως, αυτό, όπως αυτή είχε σχεδιαστεί αυτής εξ αρχής. Νομίζω λοιπόν ότι απάντησα σε όλες τις περισσότερες ερωτήσεις και σε ευχαριστώ πολύ. Uh, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις εξηγήσεις ε, που μας δώσετε και για τις ε, διαφάνειες ε, και θα θέλαμε να μας δώσετε αντίγραφα γιατί θα θέλαμε να ανεβάσουμε τις διαφάνειες στην ιστοσελίδα μας. Κύριε Βαντεκάμπ, θέλετε να ανακεφαλαιώσετε. Ίσως λοιπόν μπορείτε να μας πείτε το τι θα γίνει στο μέλλον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. να καθησυχάσω την κυρία Κορόλα. Και ο εισηγητή σα, κυρία Κορόλα, χρησιμοποιεί αυτά τα οχήματα. Και εγώ μοτοσυκλετιστή είμαι. Θα επαγρυπνήσω τόσο ώστε η νομοθεσία να μην είναι πολύ επαχθή και να μην μα πέσει στο κεφάλι. Δεύτερη παρατήρηση. Οι τροποποίησει στα μοτοποδήλατα. Αυτό είναι ένα μεγάλο, μια μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντα θα υπάρχουν Ευρωπαίοι, πάντα θα υπάρχουν νέοι που θέλουν να πειράξουν και να κάνουν πιο δυνατή τη μηχανή τους, ας πούμε, τον κινητήρα της μηχανής τους. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των νέων μας και να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι αλλαγές ε, να είναι όλο και πιο δύσκολες για να γίνουν. Φυσικά όμως οι μηχανικοί έχουν πάντα την τελευταία λέξη, κυρία Κορόλα στρέφομαι προς τον Πρόεδρο, κοιτάζω και άλλους συναδέλφους ε, για να δω τις αντιδράσεις τους. Σας ευχαριστώ όλους ε, συνάδελφοι, ευχαριστώ τους σκιώδη συναδέλφους, ευχαριστώ την Κομισιόν ε, για όλες τις απαντήσεις. Νομίζω ότι έχουμε τώρα χρήσιμα στοιχεία για αυτό το έγγραφο εργασίας, χρήσιμες προτάσεις. Προσεχώς θα γίνει μια συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών, ούτως ώστε να συμφωνήσουμε για τις διάφορες επισκέψεις που προβλέπουμε ανά την Ευρώπη. Αυτή θα είναι μια θαυμάσια πρόκληση. Ε, κυρία Ρόιλ, ε, εσείς ε, και ο κύριος Μάντος θα πάμε στην ε, Μπολόνια. Μην το ξεχνάμε. για να δούμε αυτές τις φοβερές, τα φοβερά εργοστάσια που, όπου μοντάρονται αυτές οι μηχανές. Τέλεια. Ε, δεν νομίζω ότι θα μπορέσετε να κάνετε, να καβαλήσετε τέτοιες μηχανές. Ευχαριστώ την Κομισιόν για την παρουσίαση της μελέτης αντικτύπου. Έχουμε εδώ πέρα κάποιους εκπροσώπους μοτοσυκλετιστών. Ε, ελπίζω και διάφοροι να μας παρακολουθούν από το ίντερνετ. Μόλις το συζήτησα με το, τομέα, με το τμήμα που ασχολείται με την επικοινωνία, α, πρέπει να επικοινωνήσουμε για αυτήν την πρόταση. Ελπίζω να σας έχουμε καθησυχάσει ότι και ο εισηγητής και οι υπεύθυνοι της Κομισιόν, επειδή είναι και οι ίδιοι οι μοτοσυκλετιστές, γνωρίζουν τα θέματα για τα οποία σας μιλάνε. Η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων θα γίνει στις 25 ή 26 Ιανουαρίου. Έχουμε πάρα πολλέ πληροφορίε να διαβάσουμε. Το αντίγραφο τη μελέτη αντικτύπου με πάρα πολλά στοιχεία Υπάρχει επίσης και στο διαδίκτυο αυτή η μελέτη αντικτύπου, μπορείτε να το κατεβάσετε. Ο κύριος Βάντεν Κάπ θα αρχίσει να δουλεύει την πρότασή του μετά τα Χριστούγεννα και θα τα ξαναπούμε τον Ιανουάριο. Αυτό το θέμα, δηλαδή θα συζητηθεί τον Ιανουάριο. Επίσης για το θέμα της εφαρμογής. Αυτό θα το συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση γιατί ο χρόνος έγκρισης θα σχετίζεται και με το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής. Όταν έρθετε σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους μπορείτε να μας ξαναμιλήσετε για αυτό το θέμα. Σε ευχαριστώ λοιπόν για αυτό το σημείο και τώρα περνάμε σε ένα άλλο σημείο το οποίο είναι μεγάλη σημασία για τους πολίτες επίσης και τους καταναλωτές. Αφορά την ασφάλεια των προϊόντων γενικά. Κάποια από τα προϊόντα εκπίπτουν του πεδίου εφαρμογή της, της οδηγίας, όπως ε, ε, πούμε τα ποδήλατα των παιδιών. Και αφορούν την γενική οδηγία της ασφάλειας των προϊόντων. Εκεί εντάσσονται αυτά τα προϊόντα. Η κυρία Σκαλντεμόζε κάνει μια ε, έκθεση βίας πρωτοβουλίας για την Επιτροπή μας για να δείξουμε ποια θα είναι η πολιτική μας στάση για την αναθεώρηση της οδηγίας ε, για τον έλεγχο της αγοράς και την ασφάλεια των προϊόντων. Θα δώσω την έκθεση στην κυρία Σκαλντεμόζα για να μας παρουσιάσει το κείμενό σας. Ο κύριο Κόρχολο, ο κύριο Κρόιτσμαν, η κυρία Ρούλερ, ε, δεν είναι πια εδώ, αλλά θα ξανάρθει. Ο κύριο Φόξ δεν είναι εδώ. Ο κύριο Σαλβίνη. Η κυρία Μπρίκμαν από την Κομισιόν από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων. Ο κ. Σόρου δεν είναι εδώ ακόμα. Ε, τον εκπροσωπεί κάποιο άλλος, γιατί νομίζω ότι όπου να είναι θα φτάσει. Ναι. Ε, ποιος εκπροσωπεί την ε, Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ ένα απουσία του κ. Σόρου. Α, έχουμε κάποιον από την ε, Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Ζητώ συγγνώμη, ο κύριος Σόρου και η κυρία Μάινορ βρίσκονται στο σταθμό του Λονδίνου. Ε, υπάρχει μία ε, διάσκεψη για την ε, υγεία των καταναλωτών, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να είναι στην ώρα τους εδώ. Νομίζω ότι δεν κινείται απρόσκοπτα το γύρο στα λόγω του καιρού. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Σκαλντεμόζε. Δεν έχω. Øh, Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω γιατί μας δίνετε τη δυνατότητα μέσω web streaming να αγγίξουμε ένα ευρύτερο κοινό. Να σας πω πως αναγνωρίζω ε, πως η μετάφραση της ε, έκθεση μόλις έφτασε στα χέρια σας. Ε, νομίζω χτες ή σήμερα λάβετε το κείμενο. Ελπίζω πάντως να τα έχετε διαβάσει στα αγγλικά, γιατί στα αγγλικά σας έχει σταλεί εδώ και καιρό. Να σας εξηγήσω λοιπόν εγώ για ποιο λόγο έχω παρουσιάσει αυτή την εισήγηση ίδιας πρωτοβουλίας στην Επιτροπή μας. Ε, παρόλο που υπάρχει η οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως εξακολουθεί να αποτελεί ένα ορόσημο ε, για την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Πρώτα απ' όλα, εδώ και αρκετό καιρό κάναμε την παρουσίαση μιας έκθεσης η οποία μας υπενθύμησε το ότι η κατάσταση ε, με τα μέτρα που υιοθετήσαμε το 2008 δεν είναι ιδανική και η Κομισιόν ε, έχει σκοπό να αναθεωρήσει την οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων. Έτσι λοιπόν νομίζω πως ε, λογικό θα ήταν να εξετάσουμε αυτούς τους κανόνες και να ε, δούμε αν χρειάζεται να ληφθούν μέτρα σε κάποιους κλάδους. Η δική μου γνώμη είναι πως ναι, αλλά το ζήτημα είναι πώς θέλουμε να προχωρήσει η εσωτερική αγορά και πώς θέλουμε να επανακινήσουμε και να επανεργοποιήσουμε την ε, εσωτερική αγορά. Πιστεύω πως αυτό μπορεί να γίνει με κάποιες απλές προσπάθειες και χρησιμοποιώντας τις διατάξεις που έχουμε για την γενική ασφάλεια των προϊόντων. Εάν θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά θα πρέπει να το κάνουμε μέσω κάποιων μέτρων που θα δώσουν στους καταναλωτές ε, αυτή, το, αυτή την αίσθηση ασφάλειας που τους λείπει. Ε, όμως αυτό εξαρτάται από τα μέτρα που θα λάβουμε και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Εγώ δεν θεωρώ πως η χρηματοπιστωτική κρίση αυτή τη στιγμή είναι ικανό επιχείρημα για να μην εγκρίνουμε νομοθεσία η οποία θα είναι πιο αυστηρή από την υφιστάμενη. Το σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσουμε την κρίση την οποία περνάμε αυτή τη στιγμή για να περάσουμε κάποιους αυτηρούς κανόνες, γιατί αν δώσουμε στους καταναλωτές μας μία αγορά που θα είναι ασφαλής, με ξεκάθαρους κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων, τότε οι καταναλωτές αυτοί ε, θα αγοράζουν περισσότερο. Γιατί ακούσαμε για κάποιες επικριτικές φωνές που μας είπαν ότι μην κάνετε πιο αυστηρούς κανόνες, έτσι κι αλλιώς με την κρίση η κατανάλωση έχει μειωθεί. Λοιπόν, προτάσεις. Για να εφαρμόσουμε το σύστημα παρακολούθησης της αγοράς και για να το συντονίσουμε καλύτερα, αυτά είναι τα αιτήματα που ακούμε και από τις Εθνικές Αρχές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου είναι όλοι περισσότερο συντονισμό, πιστεύω πως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα είδος ομπρέλας που θα είναι το κοινό πλαίσιο ε, για την ε, παρακολούθηση και επιτήρηση της αγοράς. Μιλάμε λοιπόν για το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα αποτελέσει τμήμα ε, της οδηγίας για την γενική ασφάλεια των προϊόντων. Άρα λοιπόν το πλαίσιο θα πρέπει να είναι κοινό και στις δύο περιπτώσεις που παρουσίασα και νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα στα κράτη-μέλη πως θα πρέπει να διαθέσουν περισσότερους πόρους οικονομικούς και ανθρώπινους στο θέμα αυτό. Θα πρέπει δηλαδή να είναι σε θέση να παρακολουθούν με αποτελεσματικό τρόπο της αγοράς. Θα πρέπει να λαμβάνουν δείγματα, να κάνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους που θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια των προϊόντων. Διαφορετικά, εάν δεν γίνονται αυτοί, οι καταναλωτές δεν θα αισθάνονται ασφαλείς. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά επιχειρήματα ε, για που συνηγορούν υπερ προτείνω, δεν θα αναφερθώ σε όλα. Νομίζω όμως πως θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την Κομισιόν να δημιουργήσει μια ε, υποχρεωτική βάση δεδομένων έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν ε, να κοινοποιούν τα ατυχήματα για παράδειγμα τα οποία έχουν διαπιστωθεί ε, έτσι ώστε να διαπιστώνεται πως κάποιο προϊόν δεν είναι σίγουρο. Δηλαδή, για τα όσα συμβαίνουν με τα διάφορα προϊόντα, καλό θα είναι να έχουμε μια κοινή βάση δεδομένων που θα έχουμε όλες τις πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό θα γνωρίζουμε καλύτερα και σε ποιους κλάδους θα πρέπει να νομοθετήσουμε μελλοντικά. Δεν θέλουμε λοιπόν να παρεμποδίσουμε την κυκλοφορία προϊόντων, αλλά πρέπει να στήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέπουν ε, τα προϊόντα τα οποία είναι λατωματικά να τα γνωρίζουμε. Αυτά τα οποία για παράδειγμα προκαλούν ατυχήματα. Ξέρουμε πως είχαμε τέτοιου είδους ατυχήματα στην Ευρώπη. Με παιδιά για παράδειγμα που πνίγηκαν, για παράδειγμα, με ε, τα λάστιχα από τα παιχνίδια με τα οποία έπαιζαν ή ε, με κορδέλες από κουρτίνες ή με κάποιον άλλο τρόπο. Μιλάμε λοιπόν για παιδάκια τα οποία πνίγηκαν με τον τρόπο αυτό. Με τα διάφορα κορδόνια που με τα οποία έπαιζαν. Λοιπόν, θα πρέπει να αποφύγουμε τέτοιου είδου ατυχήματα στο μέλλον και θα πρέπει να έχουμε πληροφορίε συγκεκριμένε για του κλάδου για του οποίου χρειάζεται περισσότερη νομοθεσία. Δεν είναι μόνο αυτό. Όταν μιλάμε για παρακολούθηση και επιτήρηση τη αγορά. Ε, υπάρχει χώρος για βελτιώσει. Αυτό που προτείνω επίση είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει αυτή την αναθεώρηση της οδηγίας για την ε, ποιότητα των προϊόντων, την ασφάλεια των προϊόντων, ε, έτσι όπως μας είχε υποσχεθεί, δεν χρειάζεται να το αφήνουμε άλλο, έφτασε η ώρα του. Και θα πρέπει να ε, ερευνήσουμε απλώς το περιεχόμενο αυτής της οδηγίας για την γενική ασφάλεια των προϊόντων, να δούμε λοιπόν σε ποια σημεία χρειάζεται να ενισχυθεί. Θεωρώ απαραίτητο να έχουμε ορισμούς πιο συγκεκριμένους, πιο σαφείς, με συγκεκριμένες απαιτήσεις για τους ε, ε, επιχειρηματίες και όλα αυτά στο νέο νομοθετικό πλαίσιο. Χρειάζεται να ακολουθήσουμε κοινού κανόνες. Και νομίζω πως ε, ακόμα και για τους κοινού κανόνες είναι απαραίτητο να αναθεωρήσουμε την οδηγία για τη γενική ασφάλεια και για παράδειγμα να σταθούμε ιδιαίτερα στους κανόνες για τη χρήση οχημάτων που δεν έχουν ενταχθεί σε αυτή, γενική, για την, σε την οδηγία για τη γενική ασφάλεια. Και βέβαια έχουμε και κάποια συγκεκριμένα θέματα τα οποία αν αναθεωρούσαμε ενδεχομένως θα καλύπταμε με καλύτερο τρόπο. Δεν χρειάζεται βέβαια συγκεκριμένους ορισμούς για, για προϊόντα που χρησιμοποιούνται από παιδιά. Νομίζω πως εκεί θα έπρεπε να έχουμε συγκεκριμένες απαιτήσει για αυτά τα προϊόντα που επαναλαμβάνω δεν είναι παιχνίδια αλλά χρησιμοποιούνται από παιδιά που λόγω χρώματος ή σχήματος είναι πολύ ελκυστικά και για τα προϊόντα αυτά νομίζω πως καλό θα ήταν να έχουμε συγκεκριμένες απαιτήσει ασφάλειας. Να, έναν ορισμό που θα καθορίζει τι, ποιο προϊόν είναι ελκυστικό για τα παιδιά. Και εκεί να έχουμε προδιαγραφές ασφάλειας. Στην τρέχουσα νομοθεσία το ίδιο προϊόν ε, ανάλογα με τον καταναλωτή που το χρησιμοποιεί μπορεί ε, αν το χρησιμοποιεί ο καταναλωτής να εμπίπτει στην οδηγία και αν το χρησιμοποιεί ε, κάποιος επαγγελματίας να μην εμπίπτει. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα κενό το οποίο εμείς πρέπει να κλείσουμε και θα μπορούμε να το κάνουμε αναθεωρώντας την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Το τελευταίο στοιχείο και αυτή είναι και η τελευταία πρόταση την οποία καταθέτω, είναι θα πρέπει οι κατασκευαστές καινοτόμων προϊόντων πριν θέσουν σε κυκλοφορία ένα προϊόν, να αναλύουν τους κινδύνους του προϊόντος αυτού. Δηλαδή, οι κουρτίνες που είπαμε προηγουμένως, ε, αυτά τα κορδόνια που μπορούν να προκαλέσουν ασφυξία, θα πρέπει όλα αυτά να καλύπτονται από το συγκεκριμένε διατάξει έτσι ώστε να φέρει ειδοποίηση ε, ασφάλεια σε αυτό το προϊόν όταν το αγοράζει κανείς. Δηλαδή ότι θα πρέπει κανείς να το χρησιμοποιήσει με προσοχή. Μια ανάλυση κινδύνου. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Τέτοιου είδου προειδοποίηση. Και αν πρόκειται για επικίνδυνο προϊόν, σήμερα με την οδηγία για την γενική ασφάλεια των προϊόντων έχουμε κάποιες διαδικασίες οι οποίες καλύπτουν αυτούς τους κινδύνους, όμως με προσωρινό τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε και εδώ την οδηγία έτσι ώστε ένα προϊόν να μην απαγορεύεται μόνο για ένα έτος, αλλά να ε, ε εξορίζεται από την εσωτερική αγορά αν δημιουργεί τέτοιου προβλήματα. Ε, νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να καλύψουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας εξηγήσει πώς μπορούμε με την ε, νέα τεχνολογία να ειχνηλατούμε την πορεία αυτών των προϊόντων. Για παράδειγμα ένα microchip ε, πώς χρησιμοποιείται. Έχουμε τις διατάξεις περί ιδιωτικού χώρου και προστασίας των ιδιωτικών δεδομένων. Οι νέες τεχνολογίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ισορροπώντας εδώ με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, με τις επιταγές της ασφάλειας. Ασφάλειας των προϊόντων. Κάτι που θα ήθελα να σχολιάσω ακόμα είναι το σύστημα RAPEX. Το οποίο είναι εξαιρετικό. Το οποίο όμως και αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί και πολλοί από τους ενδιαφερόμενους θα επιθυμούσαν να έχουν ε, πρόσβαση στα στοιχεία των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο σύστημα RAPEX. Νομίζω πως τα ασφαλή προϊόντα θα έπρεπε να περιγράφονται με διαφάνεια Άρα λοιπόν η πρόσβαση στη βάση δεδομένων των προϊόντων που καλύπτονται από τους καταλόγους RAPEX θα πρέπει να δίδονται τους πολίτες, τους καταναλωτές, έτσι ώστε να να διδαχτούμε και από τα σφάλματα των υπολείπων. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε καλύτερη ελεύθερη πρόσβαση στο RAPEX για να μπορούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε προϊόντα, για παράδειγμα, που προέρχονται από χώρες ε, Τη Ευρωπαϊκή Ένωσης γιατί ξέρουμε πώ είναι πολύ δύσκολο να έχουμε χνηλασιμότητα προϊόντων, για παράδειγμα, μέχρι τον κατασκευαστή σε περίπτωση που είναι έξω κοινοτικό, για παράδειγμα, έρχεται από την Κίνα. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε όμω τουλάχιστον για τα κοινοτικά. Τώρα, θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε και το ράπεξ για, προς κάποια κράτη με τα οποία έχουμε εμπορικέ σχέσει. Την Κίνα, επαναλαμβάνω. Ε, Μήπω πρέπει λοιπόν να αξιολογήσουμε κατά πόσο χρειάζεται αυτό για τα προϊόντα εκείνα. Γιατί η αυτών των προϊόντων δημιουργεί δυσκολίες και είναι ένας χώρος στον οποίο εμείς θα μπορούσαμε να παρέμβουμε. Πείτε με λοιπόν τι πιστεύετε, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη των σκηνόδων εισηγητών αλλά και των υπολείπων συναδέλφων. Πάντως πιστεύω πως η οδηγία χρειάζεται οπωσδήποτε αναθεώρηση και στο περιεχόμενό της και στους ορισμούς έτσι ώστε να έχουμε ένα πλαίσιο που θα κάνει τους καταναλωτές να αισθάνονται πιο ασφαλείς. Αναμφίβολα Χρειαζόμαστε να ενισχύσουμε τα συστήματα παρακολούθησης της αγοράς, γιατί οι πόροι που διαθέτουμε θα πρέπει να αυξηθούν και θα πρέπει να συντονιζόμαστε και καλύτερα μεταξύ μας. Για την ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 14 Δεκεμβρίου. Εκπνέει. Σε δύο εβδομάδες λοιπόν, δεν ε, μας λείπει χρόνος, δύο εβδομάδες έχετε στη διάθεσή σας. Και θα το περάσουμε θα το συζητήσουμε μάλλον 26-27 Ιανουαρίου εδώ στην Επιτροπή και μετά θα το ψηφίσουμε. Οπότε περιμένω τα σχόλιά σας και περιμένω και τις προτάσεις ε, και τις τροπολογίες σας. Θα ήθελα να πω δε στον πρόεδρό μας πως χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω πως και η ΙΝΤΕ και η ΙΤΕΡ θα υποβάλουν εισήγηση για τη δική μας έκθεση. Έχουμε εδώ τα μέλη αυτών των επιτροπών που στις δύο επιτροπές τις οποίες ονόμασα προηγουμένως θα ασχοληθούν με τη σύνταξη των, εκθέσεων, των εκθέσεων αυτών όπου έχουμε πάντα όλοι ως σκοπό την προστασία του καταναλωτή στην εσωτερική αγορά. Well, I wasn't uh, that we... Κοιτάξτε, εγώ δεν ενισχύστηκα παρέστα, ότι είμαστε η μόνη επιτροπή που εργάζεται για την προστασία του καταναλωτή, αλλά έθεσε ένα γενικότερο θέμα ότι θα ήταν καλύτερα να συμμετέχουν περισσότερο οι πολίτε στι εργασίε μα. Ε, και σα ευχαριστώ πολύ γιατί αυτά που μα είπατε ήταν ε, ιδιαίτερα κατανοητά, πολύ ε, επικοδομητική η εκθεσή σα και στη τελική ανάλυση περί αυτού πρόκειται. Ας πάμε τώρα στους σκιώδεις εισηγητές η κυρία Κόχαλεν, ο κύριος Κόιτσμαν, ε, ο κύριος Φόξ. Ξεκινάμε με την κυρία Κόχολα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το πάρα πολύ καλό σχέδιο έκθεσης το οποίο εξετάζει όλα τα σημαντικά θέματα. Η αποτελεσματικότητα της ε, εποπτείας ε, στην αγορά αυτό σημαίνει ότι η αγορά δεν λειτουργεί εύρυθμα σε όλα τα κράτη-μέλη. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, το να αυξηθούν οι πόροι για την εποπτεία της αγοράς, αυτό μάλλον δεν θα συμβεί στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν καλύτερα να συζητήσουμε ποιο θα είναι στο μέλλον ο ρόλο τη Επιτροπή και κατά πόσον η εποπτεία τη αγορά μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη μέσα από ενισχυμένο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, το να υπάρχει καλύτερο συντονισμό ε, ανάμεσα στι διάφορε αρχέ εποπτεία, εθνικέ και ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα βοηθήσει στο να υπάρχει καλύτερη εποπτεία. Ε, Θεωρώ λοιπόν ότι τα προϊόντα που δεν είναι αρμονισμένα ε, και όλα τα άλλα θα πρέπει ίσως να μπουν κάτω από έναν κανονισμό για την εποπτεία της αγοράς. Όσον αφορά τώρα ε, τις ε, την ασφάλεια των προϊόντων από την Κίνα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως ακριβώς αναφέρθηκε και στην γνωμοδότηση. Ε, της Επιτροπής μας. Πρέπει να βελτιωθεί η χνηλασιμότητα, αλλά και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε όλες τις επιχειρήσεις και σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων μία και μόνο λύση. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω αφορά ε, στον ορισμό των προϊόντων που είναι ελκυστικά για τα παιδιά. Νομίζω λοιπόν ότι είναι δύσκολο να βρεθεί ένας τέτοιος ορισμός και ε, πριν προκύψει ε, θα πρέπει να τον έχουμε σκεφτεί καλά. Η ασφάλεια των παιδιών είναι πολύ μεγάλη σημασία και ε, θα πρέπει να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν στην οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Να μην ξεχνάμε βέβαια και την ευθύνη των γονέων, οποτεδήποτε συζητάμε για αυτόν τον ορισμό και πώς ακριβώς αυτά τα προϊόντα πρέπει να αντιμετωπίζονται στην πράξη. Γιατί αλλιώς ε, είναι δυνατόν να υπάρξουν απρόβλεπτα εμπόδια στην δημιουργικότητα των σχεδιαστών ε, παιχνιδιών. Και ολοκληρώνοντας να κάνω και μία ερώτηση σχετικά σχετικά με την τράπεζα δεδομένων των προϊόντων αυτών. Από πού θα προέλθει αυτή η τράπεζα δεδομένων, τι θα δημοσιευθεί και τι θα υπάρξει, πώς θα συσχετιστεί αυτή η τράπεζα δεδομένων με το σύστημα RAPEX. Ο κύριος Κότσμαν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για την εποπτεία της αγοράς και στη Γερμανία παραδείγματος χάρη για μα αρμόδια για την εποπτεία της αγοράς είναι τα κρατήδια άρα δηλαδή ακόμα μεγαλύτερη κατηγοριοποίηση και το πράγμα γίνεται δύσκολο αν είναι κανείς καλά ενημερωμένος θα γνωρίζει ότι ε, τα διάφορα κρατημέλη αντιμετωπίζουν διαφορετικά την εποπτεία της αγοράς και διαφορετικά είναι και τα κονδύλια που διαθέτουν για αυτήν. Δηλαδή υπάρχουν κρατημέλη ε, τα οποία είναι χαλαρά, αν μου επιτρέπετε τον όρο, και υπάρχουν άλλα τα οποία το θέμα αυτό ε, το θεωρούν πολύ σημαντικό. Ε, οποτεδήποτε λοιπόν ε, έχω κάνει κάποια ερώτηση στον Επίτροπο για το θέμα αυτό, ε, μου έχει απαντήσει αρμόδια είναι τα κράτη-μέλη. Και αυτό δεν βοηθάει, διότι όταν τα προϊόντα έχουν φτάσει πια στα κράτη-μέλη, κατά κανόνα είναι πια πολύ αργά. Φτάνω λοιπόν στην εξή πρόταση. Μήπως να σκεφτούμε να ενισχύσουμε περισσότερο τα εξωτερικά όρια της κοινή αγοράς. Και υπάρχει ένας ε, οργανισμός, ένας θεσμός, τον γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, πρόκειται για τη Frontex. Εκεί λοιπόν τα ίδια τα κράτη-μέλη βοηθούν τα άλλα που πλήττονται ε, τα μέλη, κράτη-μέλη εκείνα όπου οι πρόσφυγες φτάνουν σε αυτά διαθαλάσσεις και με τον τρόπο αυτό δείχνουμε, επιδεικνύουμε αλληλεγγύη με άλλα κράτη που πλήττονται περισσότερο. Άρα δηλαδή και εδώ θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς. Τι σημαίνει αυτό. Έχουμε λιμάνια όπως ε, το Ρότερνταμ που ε, πραγματικά θίγονται πολύ από τα εισαγόμενα προϊόντα και ως εκ τούτου ε, θα πρέπει να δούμε λιγάκι κατά πόσον πρέπει να έχουμε κοινέ ενέργειες εποπτείας, να έχουμε τον καθορισμό λειτουργικών ε, στάνταρτ, να εκπαιδευτούν ειδικοί τελωνιακοί, να υπάρξει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 συγκέντρωση των τελευταίων επιστημονικών δεδομένων, η ενημέρωση των κρατών μελών, να διατίθενται οι απαραίτητε τεχνολογίε. Η κυρία Συγήτρια βεβαίω έθιξε κάποια από αυτά τα θέματα ε, και μίλησε και για την παροχή βοήθεια. Πρέπει να σα πω ότι με πάρα πολλέ προτάσει που καταθέσατε για την εποπτεία τη αγορά συμφωνώ. Πρόκειται για μια πολύ καλή βάση. Υπάρχουν όμω και κάποιε άλλε παρατηρήσει που αφορούν στην ασφάλεια των προϊόντων. Δεν είμαι σίγουρο για το κατά πόσον θα πρέπει να έχουμε ειδικέ προδιαγραφέ για τα παιχνίδια των παιδιών. Υπάρχει η οδηγία περί παιχνιδιών και αν υπάρχουν ελλείψεις να αντιμετωπιστούν εκεί. Τώρα, το κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει ενιαίος ορισμός, αυτό το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Μπορούμε να δοκιμάσουμε αν θέλετε, αλλά εγώ έχω πολλές αμφιβολίες. Εκείνο που δεν βρίσκουμε σημαντικό είναι να υπάρχει η ανάλυση κινδύνου κατά τη διάρκεια ε, του, του σχεδιασμού. Και πρέπει να πούμε ένα πράγμα. Δεν θα υπάρχει κανένα προϊόν στην αγορά που να είναι επικίνδυνο και επιζήμιο για τον καταναλωτή. Οι Αμερικανοί είναι πιο γενναιόδοροι, έχουν τις περίφημες ε, συλλογικές ε, ε, δίκες και όταν οποτεδήποτε ο καταναλωτής αποδεικνύει ότι έχει δίκιο, αποζημιώνεται. Αν έχουμε όμως μια υποχρεωτική ανάλυση ε, κινδύνου στη φάση της σύνταξης, κυρία Σκαλτεμόζε, αυτό θα ήταν ε, καλύτερο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι οι μεγάλες εταιρείες έχουν ε, τα λεφτά και το προσωπικό για να το κάνουν. Ε, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις θα δυσκολευόντουσαν. Το ίδιο αφορά και τα νέα τρόφιμα. Υπάρχουν ορισμένε περιοχές που πρέπει να κάνουμε αλλαγές, τροπολογίες, αλλά το πρώτο σχέδιο γενικά μου φαίνεται καλό, ειδικά για την ε, εποπτεία της αγοράς. Πρέπει να δούμε βεβαίως και τη μέθοδο που θα εφαρμόσουμε. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις ε, πιο προηγμένες τεχνολογίες, ε, τα τσιπάκια, τους μικροπροσέσορες, γιατί υπάρχουν τόσα πολλά προϊόντα που κατακλείσουν τις αγορές μας και χρειαζόμαστε ανιχνευσιμότητα σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι λοιπόν μια θαυμάσια βάση για να εργαστούμε και θα πρέπει βεβαίως ε, να συζητήσουμε και ένα-δύο σημεία που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. Αλλά συμπερασματικά ε, δεν πρέπει να αφήσουμε την ε, Επιτροπή να πει «Α, κοιτάξτε, δεν είναι δουλειά δική μου, είναι τα κράτη-μέλη που αποφασίζουν». Τα, τα κράτη-μέλη με τη σειρά τους λένε «Δεν έχουμε αρκετό προσωπικό ή δεν έχουμε αρκετά χρήματα». Ε, η Κομισιόν δηλαδή το παίζει πόντιο πιλάτο και δεν γίνεται τίποτα. Θα πρέπει να υπάρχει μια ισοτιμία α, στην εποπτεία τη αγορά. Δεν έχει κανένα νόημα να έχω μια οδηγία ενό νέο κανονισμό αν κανένα δεν τη σέβεται. Και αν οι εισαγωγεί προσπαθήσουν να παρακάμψουν του κανόνε μα, Ξέρετε ότι μπορούν να βρουν πάντα την χιλιοπτέρνα και να μπουν στην Ευρώπη. Ε, ξέρουν ότι σε κάποια κρατημέλη υπάρχει λιγότερη υποπτία. Αυτή τη στιγμή μπουν τα προϊόντα στην εσωτερική αγορά, θα είναι πολύ δύσκολο μετά να τα ξεφορτωθούμε. Αυτά τα προϊόντα έτσι, χαμηλής ποιότητας και τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπά μας. Οπότε υπάρχει εδώ μεγάλο πρόβλημα. Πρόεδρος. Ο κύριος Φόξ είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Σκάλτε Μόζε για ε, την πλήρη αυτή και σφαιρική προσέγγιση της έκθεσής της. Το αποτέλεσμα είναι μια καλή και ισορροπημένη έκθεση ενώπιόν μας. Καταρχάς, να σχολιάσω το σημείο 5, δηλαδή την ανάγκη να διαδίδουμε τις ε, βέλτιστες πρακτικές. Συμφωνώ κυρία Σκαλντεμόζε. Κάποια κράτη-μέλη έχουν πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας αγορά από κάποια άλλη και το μοίρασμα των ε, πρακτικών αυτών θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της εποπτείας και θα μειώσει και, το, φορολογικού τους φορολογικούς όλη την ενιαία αγορά. Υποστήριζω την πρόταση η Γενική Οδηγία για την Ασφάλεια των Προϊόντων με την Οδηγία για την Εποπτεία της Αγοράς να συγχωνευτούν. Ε, νομίζω ότι υπάρχει και μεγαλύτερη ομοιομορφία και μεγαλύτερη διαφάνεια. Τώρα, για τα ελκυστικά προς τα παιδιά προϊόντα. Μ' αρέσει η προσέγγιση της εισηγήτριας, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι συμφωνώ με τις δύο προλαλήσεις σας που λένε ότι θα είναι δύσκολο να το πετύχουμε αυτό από νομικής άποψης. Διερωτώ με, μήπως μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση θα ήταν να έχουμε συγκεκριμένα πρότυπα τα οποία μπορούμε να τα τροποποιήσουμε πιο εύκολα όταν χρειάζεται παρά να προσπαθήσουμε να προβούμε σε ένα νομικό ορισμό που αν χρειαστεί να το αλλάξουμε ας πούμε, α, ε, θα έχουμε τέρμονες συζητήσεις. Ούτως ή άλλως, πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να περιμένουμε την έκθεση για την κοινή δράση Για το σημείο 21, η πρόσβαση στην ε, διαθέσιμη, στη σχετική πληροφορία. Καταρχάς φαίνεται καλή ιδέα. Να ρωτήσω την εισηγήτρια, αν μπορεί να μου επιβεβαιώσει, αν έχει λάβει ε, νομικές συμβουλές από νομική υπηρεσία, για το αν υπάρχουν θέματα προστασίας των δεδομένων ή ε, εμπιστευτικά εμπορικά στοιχεία. Ή, αν δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και άρα μπορούμε να προχωρήσουμε επί τη βάση της πρότασής της για το θέμα των διαδικασιών τυποποίησης. Συμφωνώ, θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική. Απλώς αμφισβητώ το να προσθέσουμε ε, και άλλο ένα επίπεδο ε, ελέγχου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σοφό αυτό ή απλώς ε, επαυξάνουμε και την γραφειοκρατία και μεγαλώνουμε και τις προθεσμίες, προκαλούμε δηλαδή καθυστερήσεις. θα πρέπει να έχουμε πιο αποτελεσματικές διαδικασίες τυποποίηση. Αυτός είναι ο στόχος. Κύριε Πρόεδρε, Κλείνω με αυτά και ευχαριστώ την εισηγήτρια για την ε, καλή δουλειά της. Και εγώ σε ευχαριστώ κύριε Φόξ. Τώρα, ο κύριος Βάμπ και η κυρία Γκέρπχαρτ ε, είναι οι δύο βουλευτές που θέλουν να πάρουν μέρος στη συζήτηση. Ε, άλλος κανείς όχι, ο κύριος Βάμπ πρώτος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια και την κυρία Κορχόλα που είναι η σκιώδης ε, εισηγήτρια για την ε, εργόδη προσπάθειά τους και για τη συζήτηση. Όπως είπαν οι συνάδελφοι, η πρόταση που έχουμε μπροστά μας έχει καλές ιδέες. Θέλω να θέσω καταρχάς το θέμα της ανάλυσης κινδύνους ό,τι αφορά τα προϊόντα Κοιτάω το 20, 21, 22 και 23, τα σημεία αυτά στην έκθεση. Υπάρχει το σύστημα RAPEX που προσπαθεί να καλύψει αυτό το θέμα. Η κυρία Σκαλτεμόζε αναφέρθηκε στο πρόβλημα προϊόντων από την Ινδία. Δεν κοίταξα τις τελευταίες στατιστικές, το ομολογώ, αλλά άκουσα από εταιρείε ότι κάποια κρατημέλη λαμβάνουν όλο και περισσότερες αιτήσει για εισαγωγές. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν η έκθεσή σας να αξιολογήσει τις τελευταίες μελέτες RAPEX για να δούμε σε ποια κρατη έχουμε αύξηση των στατιστικών και γιατί. Γιατί υπάρχουν νέοι κίνδυνοι, πιο επικίνδυνα προϊόντα δηλαδή, ή γιατί η εποπτεία της αγοράς αρχίζει να λειτουργεί στα κράτη-μέλη. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν τόσες τόσα στοιχεία που μιλάνε για αύξηση των επικίνδυνων προϊόντων. Συμφωνώ με τον κύριο Φόξ και με τον κύριο Κρότσμαν ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτω ώστε ε, να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Το θέμα λοιπόν τη ανάλυση των κινδύνων, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα άλλο θέμα για το οποίο μίλησε επίση ο συνάδελφο κύριος Κρότσμαν αφορά στο κατά πόσον είναι δυνατόν προϊόντα τα οποία αφορούν κυρίως τα παιδιά να οριστούν και πέρα από την οδηγία για τα παιχνίδια. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Σαλμόζε γιατί από κοινού κάναμε μία προφορική ερώτηση στην Κομισιόν. Ζητήσαμε τα αποτελέσματα σχετικά με την οδηγία για τα παιχνίδια και για τις ε, τιμές ε, των ε, χημικών ουσιών. Θέλω λοιπόν να πω ότι όταν είδα την έκθεση κατάλαβα και συνεπέρανα ότι μπορεί κανείς ε, το πριόνι, το ηλεκτρικό, να το θεωρεί πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν μπορεί κανείς να το εντάξει μέσα στην οδηγία για τα παιχνίδια. Τι θέλω να πω, θέλω να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να καθορίσει κανείς το όριο. Ε, κατά τα άλλα, ε, θα ήθελα να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία που προέκυψε. Και εμείς ε, ευχαριστούμε κυρία Κέπχατ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ επίσης την κυρία Σαλδεμόζε για την, το θαυμάσιο σχέδιο έκθεσης το οποίο κατέθεσε. Είναι ένα σχέδιο έκθεσης το οποίο θίγει διάφορα θέματα τα οποία είναι πολύ μεγάλης ε, σημασίας κυρίως όσον αφορά στο θέμα της ασφάλειας προϊόντων. Πρέπει λοιπόν να πω ότι βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό που είπε ο κύριος Κρόιτσμαν. Κύριε Κρόιτσμαν, ποτέ δεν περίμενα ότι εσείς ε, θα υπερασπιζόσασταν ε, τις ε, συλλογικές ε, αγωγές. Ποτέ δεν το περίμενα αυτό. Ε, είπατε ότι τις εγκρίνετε, τις στηρίζετε και αναφέρετε και ένα επιχείρημα υπέρ αυτών. Εγώ δεν συνεπέρανα ότι γενικότερα είσαστε υπέρ των συλλογικών αγωγών, όμως αναφέρετε συγκεκριμένο επιχείρημα ισχυριζόμενος ότι η ασφάλεια των προϊόντων στις ΗΠΑ μπορεί να αντιμετωπιστεί με χαλαρότερο τρόπο γιατί ακριβώ με αυτό το σύστημα των συλλογικών αγωγών είναι δυνατόν να ασκηθεί πίεση. Αυτό ομολογώ με εντυπωσίασε συνάδελφε κύριε Χόιτσμαν και σα ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και νομίζω ότι κάπω έτσι ζωντάνεψε και η όλη συζήτηση. Κατά τα άλλα, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το θέμα των παιδιών. Και εδώ λοιπόν θα ήθελα να επενέσω ιδιαίτερα τη δουλειά της Κρίστελ, διότι η Κρίστελ στο σχέδιο της έκθεσης δεν αναφέρεται σε αυτό καθεαυτό το παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι αντιμετωπίζεται στην οδηγία περί παιχνιδιών. Ε, δεν ξέρω κατά πόσον είναι ικανοποιητική ρυθμίση. Τέλος πάντων υπάρχει εκεί μια λύση. Υπάρχουν άλλα προϊόντα τα οποία είναι κοντά στα παιδιά, που μπορεί να είναι ελκυστικά για τα παιδιά και τα οποία άλλα αυτά αντικείμενα εξαιρέθηκαν από την οδηγία περί παιχνιδιών παρότι είναι προϊόντα για τα παιδιά ακριβώς επειδή δεν μπορεί κανείς να τα να τα χαρακτηρίσει αυστηρά παιχνίδια. Αυτό λοιπόν Αυτά πρέπει να τα προσέξουμε. Και αυτό καλούμεθα να κάνουμε. Έχω λοιπόν κατά νου όχι μόνο το ηλεκτρικό πριόνι που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο γιος του κυρίου Σβάπ, αλλά έχω κατά νου ε, ένα αναπτήρα που μοιάζει με Mickey Mouse ή άλλα προϊόντα τα οποία μπορεί να είναι πολύ ελκυστικά για τα παιδιά παρότι δεν προβλέπονται για παιδιά. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε με αυτά τα προϊόντα. Γνωρίζω ότι στην οδηγία για τα παιχνίδια λύθηκαν αρκετά θέματα, όμως ε, ε ξέρουμε ε, και με το σύστημα RAPEX ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα και ότι οφείλουμε να επιληφθούμε των προβλημάτων αυτών. Όσον αφορά το RAPEX, κοιτάξτε, εγώ το κοιτάω αυτό το RAPEX ε, αρκετά συχνά γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το 80% των προϊόντων περίπου είναι παιχνίδια και ε, στο μεγαλύτερο βαθμό προέρχονται από την Κίνα. Τα περισσότερα από αυτά προέρχονται από την Κίνα. Ε, πάντως με εντυπωσίασε το ότι τα προϊόντα που δεν προέρχονται ούτε από την Κίνα ούτε από την Ασία ε, πρόκειται για προϊόντα τα οποία προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λοιπόν τίθενται ερωτήματα που έχουν σχέση με την υπευθυνότητα των επιχειρήσεων απέναντι στους πολίτες. Γιατί αυτό που κάνει το RAPEX δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ασφαλείας. Πρόκειται για προϊόντα που δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις προδιαγραφές και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Δηλαδή δεν πρόκειται μόνο για την εισαγωγή των προϊόντων αλλά πρόκειται και για προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί λοιπόν το θέμα της εποπτείας ε, της αγοράς τίθεται και πάλι τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε τέτοιου είδους προϊόντα να μην εμφανιστούν καν στην αγορά. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και κυρία Σαλντεμόζε, ε, για να μπορέσει και η να ε, συντάξει αυτή την έκθεση, άλλες πολιτικές ομάδες δήλωσαν την δήλωση αναποχή. Εγώ όμω ε, θέλησα να λάβω το λόγο γιατί ο κάθε βουλευτή είναι ελεύθερο να πει ότι νομίζει. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να συζητήσουμε το τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το σήμα ασφαλεία έτσι ώστε κάποια στιγμή ε, πράγματι το σήμα αυτό να είναι αξιόπιστο. Right. Does anyone else, um, anybody else είναι πολύ ε, δύσκολο ε, να ε, αγνοήσει κανείς τον κύριο Κρότσμαν και τον κύριο Γκέπχαρτ γιατί παρακολουθούν τα θέματα πολύ κοντά εκ του Επιτρέψτε μου να κάνω εγώ ένα σχόλιο, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να σημειώσουμε τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Όπως ξέρετε πολύ καλά, είχα το ε, προνόμιο να με καλέσουν σε αυτή την τριμερή συνάντηση πρόσφατα και θα ακούσετε και μια έκθεση που ε, θα σας ε, παρουσιάσω. Ένα ανακοινοθέν θα είναι. Θεωρώ ότι έχει βελτιωθεί κατά πολύ η σχέση και ίσως μπορούμε να ενθαρρύνουμε λιγάκι τις εξελίξεις, κυρίως την ανταλλαγή πληροφοριών για την οποία μιλήσατε. Και ίσως μπορούμε να προσθέσουμε και κάτι άλλο. Είχαμε ένα σεμινάριο στο οποίο επίσης συμμετείχα και στο σεμινάριο εκεί έγινε κυρίως λόγος ε, για τον σχεδιασμό προϊόντων. Ε, αναφερόταν σε κινέζικες εταιρείες. Αυτό είναι ένα πολύ ευρύ θέμα, ε, το θέμα των κινέζικων προϊόντων. Βεβαίως και πρέπει κανείς να ξεκινήσει με τον σχεδιασμό, αργότερα με τον έλεγχο ποιότητα και την κατασκευή. Τα, οι ευρωπαϊκές εταιρείε που έχουν προϊόντα που τα κατασκευάζουν στην Κίνα πρέπει να εξασφαλίζουν μια ασφαλή αλυσίδα τροφοδοσίας και αυτά είναι θέματα που συζητήσαμε στο σεμινάριο που σας ανέφερα. Υπάρχουν ε, σχέσεις ε, και με την Επιτροπή των ΗΠΑ που ασχολείται με την προστασία του καταναλωτή και πρέπει να το αναφέρουμε. Ο πρόεδρος αυτής της Επιτροπής είναι πρόεδρος η γυναίκα, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτά τα θέματα. Νομίζω λοιπόν ότι οι συνάδελφοι από την Επιτροπή ίσως μπορούν εκείνοι να αναφέρουν την άποψή τους. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Μπρίνκμαν και θα ακολουθήσει ο κύριος Βαντερτσέκ. Η κυρία Μπρίνκμαν παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για την εποπτεία της αγοράς θα να πω δύο λόγια. Ο Γενικός Διευθυντής μας είναι υπεύθυνο για, το, ε, για τον κανονισμό 765 για την εποπτεία της αγοράς. Καλωσορίζουμε την έκθεση που ετοίμασε η κυρία Σκαντεμόζε. Θεωρούμε ότι είναι μια θαυμάσια έκθεση που περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα και θετικά στοιχεία και προτάσεις για την καλύτερη εφαρμογή της εποπτείας της αγοράς και δείχνει και πώς μπορούμε να συντονίσουμε καλύτερα τις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς. Είναι μία δραστηριότητα των εθνικών αρχών καταρχήν, αλλά η Κομισιόν έχει ένα σημαντικό ρόλο ως προς το συντονισμό των δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό. Σας διαβεβαιώνουμε ότι το ρόλο αυτού του συντονισμού τον ε, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά και είμαστε πολύ ενεργοί και δραστήριοι. Ε, συμφωνούμε με την πρότασή σας για βελτίωση της ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και κάποιες κοινέ ε, δραστηριότητες επίσης. Μας άρεσε αυτό το κομμάτι, γιατί ακριβώς αυτά κάνουμε και εμείς τώρα σε ό,τι αφορά την εποπτεία της αγοράς με, την αντίστοιχη αρχ... με τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Τα κράτη-μέλη ζήτησαν μάλιστα από την Κομισιόν να δραστηριοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν την ανάγκη για συντονισμό. Ο συντονισμός ε, σημαίνει συντονισμό σε εθνικό επίπεδο των αρχών ε, εποπτείας αγοράς αλλά και μεταξύ των αρχών εποπτείας αγοράς των κρατών μελών και μεταξύ των αρχών αυτών εποπτείας αγοράς και των τελωνιακών αρχών. Όλα αυτά σημαίνει συνεργασία, κοινά εργαλεία, συντονισμός και χρήση των εργαλείων μάλιστα με τον ίδιο τρόπο. Γίνονται πάρα πολλά. Υπάρχει μια πυρετόδης δραστηριότητα και θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Υποστηρίζω όλα τα συμπεράσματά σας για την εποπτεία της αγοράς και αυτό που ζητάτε για ένα πιο ενιαίο νομικό πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς. Πιστεύουμε ότι είναι ενδιαφέρουσα ιδέα. Την καλωσορίζουμε. Εμείς τουλάχιστον θεωρούμε ότι είναι ένα χρήσιμο βήμα για να εξασφαλίσουμε την συνεπή εφαρμογή. Ακριβώς αυτό ζητάνε οι πάντες. Οι έμποροι, οι οικονομικοί φορείς, οι καταναλωτές, τα κράτη-μέλη. Είναι θαυμάσια η πρόταση και ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Καλησπέρα. Και εγώ ευχαριστώ την εισηγήτρια που προετοίμασε αυτή την θαυμάσια έκθεση. Συμφωνώ με την προλαλή σας από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συνέπεια σε ό,τι αφορά τις δομές των, της αγοράς. Συνεργαζόμαστε με, τα, με τους βουλευτές αυτής της Επιτροπής και προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη όλες τις χρήσιμες ιδέες για την αναθεώρηση της Γενικής Οδηγίας για την Ασφάλεια των Προϊόντων. Και θα προσπαθήσουμε ε, να τα λάβουμε υπόψη μας αυτά και στην πρόταση που θα κάνουμε και στην μελέτη αντικτύπου. Ωραία, ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Η συγγήτρια τώρα θέλει να κλείσει τη συζήτηση. Μας δώσατε το χρονοδιάγραμμα, αλλά πέστε μας. Οτιδήποτε άλλο θέλετε να πείτε. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις αυτές. Θα ήθελα καταρχήν να σχολιάσω πως τα θέματα αυτά τα έχουμε ήδη συζητήσει μεταξύ μας και εκπλήσωμε που κάποιοι, πελάτε, που κάποιοι με συγχωρείτε συνάδελφοι δεν καλύπτουν από όσα είπαμε για τα προϊόντα τα οποία είναι ελκυστικά για τα παιδιά. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα σημεία που πιο πολλές δυσκολίες προκαλεί. Εγώ σημείωσα τα σχόλιά σας και νομίζω ότι μέχρι τις 14 μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες τις οποίες θα συζητήσουμε μετά. Και ελπίζω πως θα καταλήξουμε στις καλύτερες δυνατόν λύσεις. Για τον κύριο Φόξ και τα όσα είπε για το σημείο 21, Πρέπει να σας πω πως εγώ δεν ζήτησα από την νομική υπηρεσία να, να γνωμοδοτήσει για το κατά πόσο είναι ορθή η πρότασή μου ή όχι. Πρόκειται για ε, έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Πιστεύω λοιπόν πως αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ε, δεν ξέρω τι θα μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με ποια βάση. Αν κάποια στιγμή αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια έκθεση, τότε θα πρέπει να καταλήξει σε ένα σχήμα το οποίο θα έχει το σωστό νομικό πλαίσιο. Αργότερα μπορούμε λοιπόν να δούμε τις εφαρμοστικές λεπτομέρειες και το κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί για τόσα είπε η κυρία Κόρχολα. Νομίζω πως αν δημιουργηθεί αυτή η βάση δεδομένων, αυτό μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη είναι να ορίσουν ε, στοιχεία, δεδομένα ή ατυχήματα ή συμβάντα τα οποία θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τεχνικά το πώς θα γίνει αυτό, ας το δούμε σε εθνική ε, διάσταση. Πρέπει να σας πω, στο εθνικό επίπεδο υπάρχουν πάρα πολλοί οδοί επικοινωνίας και νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε από εκεί τις βέλτιστες πρακτικές. Τώρα για την κοινή αγορά που έχουμε, να σας πω πως τουλάχιστον για τα επικίνδυνα προϊόντα υπάρχει αυτό που ζητάμε. Ξέρουμε πού είναι ο κίνδυνος και μπορούμε να προστατευτούμε. Εκεί λοιπόν λειτουργεί. Αυτό με το οποίο ικανοποιούμε είναι ότι βλέπω που συμφωνείτε σε γενικές γραμμές με την πρότασή μου και αυτά με τα οποία έχετε διαφωνίες είναι ίσως ίσονος σημασίας και όλα αυτά θα συνεισφέρουν στις προσπάθειες που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν θα αποφασίσει να αναθεωρήσει το κείμενο της οδηγίας. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε λοιπόν και την απόκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και της εισηγήτριας για, το... για την έκθεση αυτή και για το ποιο λόγο αποφασίσαμε να προχωρήσουμε. Ωραία λοιπόν, μας δώσατε το χρονοδιάγραμμα, πρώτα τροπολογίες και περαιτέρω συζήτηση τον Ιανουάριο. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο της σας είναι η πρώτη γνωμοδότηση Κρότσμαν σήμερα. Ο κύριος Κρότσμαν έχει περάσει πραγματικά δύσκολο απόγευμα και αν κατάλαβα καλά είστε συντονιστής και για τους ε, φιλελεύθερους. Είναι αλήθεια. Ωραία. Συγχαρητήρια λοιπόν ε, και για τον δραστήριο τρόπο με τον οποίο προωθείτε αυτές τις εκθέσεις. Η πρώτη λοιπόν είναι η βιομηχανική πολιτική για την παγκοσμιοποιημένη εποχή. Αυτό είναι ο τίτλος της έκθεσης που μας υπέβαλε ο κύριος Ταζανή όταν είστε στην Επιτροπή μας πριν από δύο εβδομάδες. Χαίρομαι λοιπόν που μπορώ να σας δώσω το λόγο για να παρουσιάσετε και εσείς την, την έκθεσή σας. Πρόεδρε, θα προτάξω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, η γερμανική μετάφραση είναι κάκιστη. Ε, υπάρχουν θέματα, στοιχεία που είναι λάθος. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς θα μεριμνήσουμε να διορθωθεί. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο. Προσπάθησα ότι υπάρχει στην έκθεση Λάγκε από την Επιτροπή Βιομηχανίας να μην τα επαναλάβω εδώ. Δηλαδή προσπάθησα να έχω περισσότερο μία προσθήκη και από ό,τι είδα έχουν κατατεθεί τροπολογίες τις οποίες μπορώ να δεχτώ ε, Κάποιες άλλες πρέπει να τις απορρίψουμε. Επιτρέψτε μου να κάνω μερικές ε, παρατηρήσεις. Η δική μου η πρόταση σας έχει κατατεθεί εγώ υπογράμμισα ότι η κοινωνική οικονομία της αγοράς αποδείχθηκε κάτι το ιδιαίτερα επιτυχημένο στη Γερμανία και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε οποτεδήποτε σκεπτόμεθα βιομηχανική πολιτική. Χρειαζόμαστε μια ανταγωνιστική, βιώσιμη πολιτική βιομηχανίας, μια πολιτική η οποία να μπορεί να εφαρμοστεί στην Ευρώπη γιατί με τον τρόπο αυτό θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, θα διατηρήσουμε άλλες και με θα μπορέσουμε να ε, προσφέρουμε ευημερία στους πολίτες της Ευρώπης. Αυτό που είναι καθοριστική σημασία είναι να ισχύει το πλαίσιο. Χρειαζόμαστε εναρμόνιση που να βελτιώνει την απόδοση, ε, χρειαζόμαστε εξοικονόμηση πόρων, μεγαλύτερη αποδηματικότητα, περισσότερη οικονομία, η οποία όμως θα πρέπει να υφίσταται και μεγαλύτερη εποπτεία. Χρειαζόμαστε επίσης και νομίζω αυτό το λέω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί επανειλημμένα αναφέρεται ότι πρόκειται για τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι οι υπεργολάβοι, είναι οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες κρατάνε στη ζωή τις μεγάλες επιχειρήσεις με τα καινοτόμα προϊόντα τους, με τα φτηνά προσιτά ως προς το κόστος προϊόντα τους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν την ευκαιρία να επιζήσουν και να μην τις επιβαρύνουμε με γραφειοκρατία σε περίπτωση που παρουσιάζουν καινοτόμα προϊόντα. Χρειαζόμαστε λοιπόν φιλικότητα προς τις καινοτομίε και χρειαζόμαστε και ένα ουδέτερο πλαίσιο όσον αφορά τις καινοτομίε. Να φέρω κάτι συγκεκριμένο. Σήμερα όλοι μιλάνε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και είναι τελείως διαφορετικό το ε, να έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Κίνα γιατί εκεί θα μιλάμε ε, κυρίως για αυτοκίνητα που θα χρησιμοποιούν μπαταρίες ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Αμερική όπου οι άνθρωποι χρειάζονται 2-3 ώρες για να πάνε στην ε, δουλειά τους. Εκεί λοιπόν ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία δεν θα σημαίνει δεν θα χρησιμοποιηθούν σχεδόν καθόλου γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλες δυνατότητες θα πρέπει ίσως ε, εκεί ε, να χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητα με δίζελ και με βενζίνη. Άρα δηλαδή χρειαζόμαστε ε, αυτοκίνητα που να είναι περισσότερο ουδέτερα ως προς την όθησή τους γιατί θα πρέπει να μεριμνήσουμε, να μην ε, διασπαθίζουμε τους πόρους. Η κοινωνική εταίρη. Η κοινωνική εταίρη θεωρώ ότι ενδείκνυνται κυρίως για να ε, κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές λόγω της οικονομικής κρίσης. Αυτό το ξεχνάμε πολύ συχνά. Παραδείγματος χάρη στη Γερμανία ε, έχουμε τους, ε, τις συλλόγες εργοδοτών. Εκεί υπάρχουν πολύ καλές σχέσεις και τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τους κοινωνικούς εταίρους. Μόνο έτσι μπορέσαμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Στη Γερμανία υπήρξαν πάρα πολλά εργαλεία που ήταν επιτυχημένα. Η μερική απασχόληση αυτό κατέστη δυνατόν μόνο λόγω της συνεργασίας των κοινωνικών κοινωνικών εταίρων. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό οι ε, κοινωνικοί εταίροι να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση γιατί οι κρατικές επεμβάσεις μπορούν ίσως να αμβλύνουν τις επιπτώσεις αλλά αν δεν υπάρξει η συνεργασία των κοινωνικών εταίρων δεν είναι δυνατόν να ξεπεραστούν οι κρίσεις. Επίσης οφείλουμε να μεριμνήσουμε έτσι ώστε η ευρωπαϊκή βιομηχανία να μην βρεθεί σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα ε, δεν είναι σωστό να έχουμε το βλέμμα στραμμένο μόνο στην Ευρώπη και επειδή παραδείγματο χάρη η γερμανική βιομηχανία εξάγει το 60% των προϊόντων της Ευρώπη να θεωρούμε ότι αυτό αρκεί. Χρειαζόμαστε προϊόντα τα οποία να είναι ανταγωνιστικά στην παγκόσμια αγορά και αυτές ε, ήταν οι προτάσεις ε, που καταθέσαμε εμείς ως Επιτροπή και καταθέτουμε εμείς ως Επιτροπή Κοινής Αγοράς εν είδη προσθήκης στην έκθεση Λάγκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, όσον αφορά τους ε, η, κυρία ε, θα μιλήσει εκ μέρους του συναδέλφου της, που δεν είναι παρόν. And, um, uh, Mr. Jouvin, sorry, Mr. Κύριο Ζουβά, ο κύριος κυρία Ρούλη δεν είναι εδώ. Κανένας άλλος δεν είναι εδώ. Α ξεκινήσουμε πρώτα από όλους με την κυρία Γκέπχαρτ και μετά με τον κύριο Ζουβά. Πολύ ωραία. Είχα την εντύπωση ότι θα ξεκινήσει ο συνάδελφός μου. Εντάξει, τέλος πάντων, ας ξεκινήσω εγώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κρόιτσμαν για την έκθεσή σας. Εγώ την έκθεσή σας δεν τη διάβασα στα γερμανικά, τη διάβασα στα γαλλικά. Ε, κατόπιν τούτου δεν ξέρω αν η μετάφραση που διάβασα είναι καλή ή όχι. Ε, τέλος πάντων ε, θεωρώ ότι είναι καλή. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου του κυρίου Κορέαντε Κάμπο, ο οποίο δεν μπόρεσε να έρθει, ο οποίο όμω έχει καταθέσει μια σειρά τροπολογιών, ε, τροπολογίε ε, από κοινού και με τον σκιώδη συγκητή του ΕΛΚ. Δεν θα εκπλαγείτε λοιπόν για το ότι εμεί βεβαίω δεν συμφωνούμε απόλυτα με τη δική σα την πολιτική γραμμή, γιατί ε, το δικό σα το κείμενο διακατέχεται από φιλελεύθερα συστήματα που εμεί δεν τα συμμεριζόμεθα απόλυτα. Ναι, με στην κοινωνική οικονομία της αγοράς, λέτε την αναφέρετε βέβαια, αυτά όμως που παρατίθενται στο κείμενό σας δεν έχουν σχέση με την κοινωνική οικονομία της αγοράς, αλλά με την ακρεφνή οικονομία της αγοράς και αυτό εμάς μας ενοχλεί. Γι' αυτό λοιπόν εμάς μας, ε, είναι πολύ δύσκολο να δεχτούμε το κείμενο ως έχει. Κατά τα άλλα υπάρχει μια τροπολογία ε, για την οποία θεωρώ ότι μπορείτε να τη δεχθείτε για μας δεν πρόκειται μόνο περί ανταγωνισμού όσον αφορά την αγορά, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την παγκοσμιοποίηση. Θα πρέπει αυτή να σχεδιάζεται και με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και όταν μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη δεν εννοούμε προϊόντα τα οποία να είναι βιώσιμα, βιομηχανικά προϊόντα που να είναι βιώσιμα από πλευράς ε, οικολογικής ε, ε, οικογελογικού σχεδιασμού εννοούμε πάρα πολλά περισσότερα ε, μια ευρύτερη προσέγγιση και όχι μια αμυγός οικονομική. Κατά τα άλλα υπάρχει και μια τροπολογία των κυρίων Κορέα και Άλμπερτ στην οποία τροπολογία αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική και λέμε ότι θα πρέπει αυτή να εστιάζεται σε τέτοια προϊόντα που πραγματικά είναι χρήσιμα για τον άνθρωπο. Να μην είναι μόνο χρήσιμα για τη βιομηχανία αλλά και για τον άνθρωπο. Αναφέρονται τα προγράμματα Galileo, η TGMS ως παραδείγματα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί εκεί έχουν όφελος και οι πολίτες εάν τελικά συνεχιστούν αυτά τα προγράμματα. Και πρόκειται, αν θέλετε, για ένα είδος ευρωπαϊκής μέρημνας, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω έτσι αυτόν τον ε, απλοϊκό όρο. Κατά τα άλλα, εσείς λέτε ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να εισακούνται. Βεβαίως και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, όμως ε, το ότι λέτε ότι θα πρέπει να εισακούνται και μόνο εκείνοι μπορούν να δημιουργήσουν τους κανόνες του παιχνιδιού έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την κρίση που αντιμετωπίζουμε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Εγώ εδώ διαφωνώ μαζί σας και βεβαίως και ο κύριος Κοροντεκάμπος πόσο μάλλον η δική μου η πολιτική ομάδα δεν συμφωνώ μαζί σας ότι ε, τα κράτη δεν πρέπει να επεμβαίνουν. Κάθε άλλος. Η κρίση απέδειξε το αντίθετο. Εκεί όπου λειτουργήσαν οι δυνάμεις απορρίθμισης, εκεί η κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην οξύτερη μορφή της. Άρα δηλαδή στον τομέα αυτό χρειαζόμαστε ξεκάθαρους κανόνες προφανώς και στην βιομηχανική πολιτική. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που δεν σα έδωσα την πρώτη θέση, μια και προέρχεστε από την πιο μεγάλη πολιτική ομάδα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ζητώ συγγνώμη. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη τον ε, κύριο Αμπάτ που είχε άλλε υποχρεώσει, αλλά μαζί δουλέψαμε για το θέμα, το οποίο εκείνο γνωρίζει πολύ καλά. Καταρχά, ε, επί μακρόν, ο όρο βιομηχανία ήταν ε, μια προσβολή στην πολιτική. Ήταν προσβλητικό όρο. Δηλαδή, ο τρόπο ανάπτυξη των μοντέρνων χωρών όπω οι χώρε μα θεωρείται ότι θα πρέπει να περάσει μόνο μέσω της ανάπτυξης των υπηρεσιών. Τώρα όμως που έφτασε η κρίση, ε, διαπιστώσαμε ότι είμαστε τυχεροί που κρατήσαμε βιομηχανίες, κάποιες βιομηχανίες στην Ευρώπη και συνειδητοποίησαμε ότι πρέπει να αναπτυχθούν αυτές οι βιομηχανίες. Γιατί? Για προφανείς λόγους. Ε, γιατί προάγουν την καινοτομία. Ε, το είπατε και θα το πούμε, θα το πούμε και στις τροπολογίες. Γιατί προωθούν τις θέσεις απασχόλησης. Γιατί αυτή τη στιγμή μια βιομηχανία έχει βγει από την ε, Ένωση, δεν ξαναγυρνάει. Χάνεται η τεχνογνωσία. Και η απώλεια αυτής της τεχνογνωσίας ε, σημαίνει ότι κυδεύουμε μια οικονομική δραστηριότητα. Μου κάνει εντύπωση το ξέρω, θα κάνει διαφορετική εντύπωση στους Γερμανούς. Αλλά εμείς στη Γαλλία φτιάχνουμε ακόμα πυρηνικά εργοστάσια. Πριν από 30 χρόνια, ναι, ναι, καταλαβαίνω την αντίδρασή σας. Πριν από 30 χρόνια η αγορά ήταν πάρα πολύ μεγάλη και κατασκευάζονταν πολλά πυρηνικά εργοστάσια. Η αγορά όμως έπαθε καθίζηση και αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε μόνο ένα πυρηνικό εργοστάσιο στην Ορμανδία, στη Γαλλία. Ε, δεν μπορέσαμε να κατασκευάσουμε ε, ούτε ένα εργοστάσιο δηλαδή, ενώ πριν από 20 χρόνια ε, είχαμε πολλά τέτοια πυρηνικά εργοστάσια που ε, τα χτίζαμε παράλληλα. Δεν σα το λέω για να σα πειράξω τώρα αυτό το θέμα των πυρηνικών εργοστασίων, αλλά θέλω να σα πω ότι σε όλη την, σε όλο το βιομηχανικό κλάδο χάνουμε τεχνογνωσία. Εδώ μπαίνει και το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της, ε, των τεχνητών. Θέλω να μιλήσω επίση για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Ξέρουμε τι δυσκολίε ε, που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσουμε το θέμα των διπλωμάτων αυτών. σω μέσω αυτού του κειμένου θα μπορούσαμε να προτείνουμε στην Κομισιόν να προχωρήσει με την ε, προνομιούχο εταιρική σχέση. Οι χώρες δηλαδή που θέλουν να προχωρήσουν, να προχωρήσουν και οι υπόλοιποι ας ακολουθήσουν όταν επιθυμούν. Ας δείξουμε ρεαλισμό. Αυτό είναι η Ευρώπη στο κάτω-κάτω. Πριν να τελειώσω, θα ήθελα να πω ένα σημείο, Πρόεδρε. Ε, η εσωτερική αγορά είναι η οικονομική δύναμη και ισχύ τη Ευρώπη. Είναι μια αγορά για του Ευρωπαίου αλλά παράλληλα είναι και ένα εργαλείο κατάκτηση ή αντίσταση στον εξωτερικό κόσμο. Για αυτού αυτού του δύο λόγου. Α μην είμαστε αφελεί. Νομίζω ότι επί πολύ χρόνο δείξαμε αφέλεια στι συναλλαγέ που είχαμε με του διεθνεί μα εταίρου, σε εμπορικέ συναλλαγέ, πολύ συχνά δεν προωθούμε την αμοιβαιότητα, για να καταπολεμήσουμε την μετεγκατάσταση που είναι η μάστιγα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, για να την καταπολεμήσουμε, δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να πούμε ότι θέλουμε οι ανταλλαγές βιομηχανικών αγαθών να, γίνεται, να γίνονται επί τη βάση της αμοιβαιότητας. Όταν αγοράζουμε ένα αγαθό το οποίο φέρνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα βιομηχανικό αγαθό, το κάνουμε γιατί θεωρούμε ότι ψεύεται κάποια περιβαλλοντικά κριτήρια, υγειονομικά κριτήρια, αλλά και κοινωνικά κριτήρια. Ε, ο κόσμος δεν βασίζεται στην αγάπη και στα συναισθήματα, ε, βασίζεται και στον ανταγωνισμό. Ο κόσμος αυτός χαρακτηρίζεται από ανταγωνισμό. Δεν θέλω να μου πείτε τώρα ότι προωθώ τον ε, προστατευτισμό. Δεν θέλω να με κάψετε στην πυρά για αυτά που λέω, αλλά θέλω να πω ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι αφελής. Θα πρέπει να μπορεί να προστατεύει τη βιομηχανία της και να αντισταθεί στην τάση των μετεγκαταστάσεων. Ευχαριστώ κύριε Ζουβά. Ένα-δύο σχόλια, μια, έχουμε λίγο, μια και έχουμε λίγο χρόνο. Με αυτές τις νομοδοτήσεις χρήσιμο είναι να δούμε πού μπορούμε χάρη σε αυτές να προσθέσουμε κάποια προστιθέμενη αξία. Είπατε στον κύριο Κρόιτσμαν ε, αυτά που είπατε ε, για τις δημόσιες αρχές και πώς μπορούν να βοηθήσουν ε, στην αποδοχή των νέων τεχνολογιών. Η σημασία των κρατικών προμηθειών στην ε, πρόθεση της καινοτόμας βιομηχανίας δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε και κάτι πιο συγκεκριμένο για αυτό το σημείο. Ε, το... Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στο έργο που κάνει αυτή η Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν μέσω της ομάδας μου να σας ε, προτείνω μια τροπολογία για αυτό το σημείο. Επίσης για αυτό που είπε ο κ. Ζουβά. Τα συστήματα και οι υποδομές που χρειάζονται για να υποστηρίξουμε μια ε, ισχυρή οικονομία που βασίζεται στη βιομηχανία. Υπάρχουν πολλά θέματα εδώ τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργία της παγκόσμιας αγοράς και της εσωτερικής αγοράς. Το πρώτο είναι οι, τα διαθέσιμα, οι διαθέσιμες πρώτες Υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες με πολύ συγκεκριμένες πρώτες που είναι πολύ σημαντικές για κάποιες κατηγορίες προϊόντος, παράδειγμα χάρη ψηφιακών προϊόντων. Επίσης υπάρχουν δυσκολίες με κάποια μη σιδηρούχα μέταλλα. Παραδείγματο χάρη για την αεροναυπηγική και για άλλου τομεί όμω. Ε, αξίζει να το τονίσουμε αυτό. Ε, για να συνεισφέρουμε κι εμεί έτσι. Επίση όμω θέλω να εστιάσουμε και στι δυσκολίε που πρέπει να επιλύσουμε λόγω ανεπαρκειών σε κάποια νομοθετήματα για το περιβάλλον, όπως το χάρη την ανακύκλωση. Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες ακόμα ε, για το πώς θα μεταφέρουμε ε, τα απόβλητα, πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα αξιοποιήσουμε το καλό, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον της βιομηχανίας αυτό. Ε, ειδικά στο βαθμό που έχουμε περιορισμούς στα διαθέσιμα, στη διαθέσιμη Παραδείγματο χάρη, αλουμίνιο φερρυπίν. Και το αναφέρω γιατί ε, την περασμένη εβδομάδα ήμουν σε ένα συνέδριο για το αλουμίνιο. Είναι ένα ανακυκλώσιμο υλικό το αλουμίνιο και στην ε, αεροναυπηγική χρησιμοποιούν ε, κατά 80% ε, το αλουμίνιο για να φτιάξουν ελαφρά υλικά. το αλουμίνιο είναι ανακυκλώσιμο, πρέπει να το πούμε. Είναι ένας νέος τρόπος οργάνωσης για να στηρίξουμε τη βιομηχανία. Νομίζω ότι η μεταφορά των αποβλήτων, ο κύκλος ζωής τους, ε, αυτό συνδέεται πάρα πολύ ε, με τη βιομηχανία. Ε, μην ξεχνάμε ότι η βιομηχανική παραγωγή, η βιομηχανική διαδικασία είναι κυκλική. Ε, Χθε ήμουν σε μια συνάντηση με τον κύριο Ποτότσνικ. Γνωρίζει αυτά τα θέματα ε, και νομίζω ότι θα τον βοηθήσουν αυτές οι απόψεις. Ε, μιλήσατε επίσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε κάθε βιομηχανία, σε κάθε βιομηχανικό κλάδο υπάρχει μια μακρά λυσίδα ε, προμηθευτών. Ε, ξεκινάμε από την προφορά ε, πρώτων υλών, πάμε προς μεγαλύτερες, μεγαλύτερους ενδιαμέσους και τελικά φτάνουμε στον τελικό αποδέκτη. Πιο ποιοτική προσφορά είναι σημαντική για να κρατήσουμε ζωντανή την κατασκευαστική, τη βιομηχανία εν γέννη στην Ευρώπη. Η ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να επωφεληθούν από την ενιαία αγορά, να συνεργαστούν, ε, μπορεί να οδηγεί σε προϊόντα ε, προσθέμενης αξίας. Αυτό σημαίνει διασυνοριακή συνεργασία, σημαίνει αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς Ε, δεν έχει νόημα να περιορίσουμε και να δημιουργήσουμε ασφυξία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορούν να αναπτυχθούν πέρα από τη χώρα τους. Νομίζω ότι αυτή είναι η προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει η Επιτροπή μας. Ε, σας, δίνω αυτές τις, σας προτείνω αυτές τις ε, σκέψεις για να τις ε, χρησιμοποιήσετε. Άλλος κανείς θέλει να μιλήσει. Καταρχάς να δώσω το λόγο στην Κομισιόν και μετά ο εισηγητής θα ολοκληρώσει. Ο Κρις Άλαν ε, θα μιλήσει για τις βιομηχανικές πολιτικές, ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων. Ε, μπορεί να σχολιάσει τα όσα άκουσε και να μας ενημερώσει για την πρόοδο που έχει κάνει ε, η Κομισιόν με την πρωτοβουλία της. Ευχαριστώ πολύ Μάλκομ και σας ευχαριστώ πολύ που μας δώσατε το λόγο. Εμείς χαιρετίζουμε το γεγονός πως η δική σας Επιτροπή ε, συνεισφέρει με τόσο ενεργό τρόπο στην έκθεση αυτή για τη βιομηχανική πολιτική και το θεωρούμε εξαιρετικά ικανοποιητικό. Πρέπει να σας πω πως οι προτάσεις που γίνονται σε γενικές γραμμές, όσες είδα και η συζήτηση την οποία παρακολούθησα εδώ, μου δημιουργούν την εντύπωση πως κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Άρα λοιπόν ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τα όσα έχουμε στο δικό μας, στη δική μας ανακοίνωση και τα όσα βρίσκονται υπό συζήτηση στο Συμβούλιο Ανταγωνισμού και εννοώ βέβαια τα συμπεράσματα τα οποία θα εγκριθούν 10 Δεκεμβρίου αν δεν κάνω λάθος. Έχω δύο-τρία σημεία ε, τα οποία θα ήθελα να σχολιάσω. Καταρχήν η ανακοίνωση αυτή, όπως είπε ο κύριος Ζουβά, είναι σημαντική Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά μετά από πολύ μεγάλο διάστημα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει το ρόλο της βιομηχανίας με τόσο θετικό τρόπο. Λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, πια θεωρείται η βιομηχανία ως βασικός παίκτη στο μοντέλο, το αναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας μας και κυρίως η παραγωγικότητα της βιομηχανίας ε, είναι το στοιχείο που μας απασχολεί. Η βιομηχανική παραγωγή είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν πριν από 20-30 χρόνια και αυτή η αύξηση της ε, βιομηχανικής επεξεργασίας και κατεργασίας οδηγεί σε αύξηση της ζήτηση των υπηρεσιών, των θέσεων απασχόλησης στις ε, υπηρεσίες, αλλά και, στις, ε, αλλά και αύξηση της κατανάλωσης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το αναγνωρίσουν. Όμως τούτου λεχθέντος θα πρέπει να δούμε και το πού η Επιτροπή σας θα μπορούσε να παίξει ρόλο στη διαδικασία αυτή. Εμείς καλωσορίζουμε τις προτάσεις που έκανε ο Πρόεδρος για, τα, για τις πρώτες ύλες, ακατέργαστα υλικά, για τις δημόσιες ε, προμήθειες και για τα απόλυτα. Είναι θέματα τα οποία είναι σημαντικά και όπου εσείς είσαστε μάλλον πιο εξειδικευμένοι. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλη κλάδη στους οποίους ενδεχομένως θα μπορούσατε να εξετάσετε το κατά πόσο θα μπορούσατε να προσθέσετε κάτι επιπλέον. Εγώ θα αναφερόμουν σε, σε τρία κυρίως θέματα, τα οποία για μας έχουν γίνει πιο σημαντικά. Καταρχήν, καινοτομία. Εσείς αναφερθήκατε στην τεχνολογία εχμής και στο γεγονός πως αυτή η τεχνολογία είναι απαραίτητη. Εμείς χαιρετίζουμε την ιδέα πως οι δημόσιες αρχές θα πρέπει ε, να συνηγορούν υπέρ της αποδοχής και χρήσης από, το δημόσιο των νέων τεχνολογιών με όλες τις εφαρμογές τους, αλλά αυτό το οποίο διαπιστώνουμε στις συζητήσεις που ε, κάνουμε στην ομάδα υψηλού επίπεδου είναι πως υπάρχει μια πραγματική ανάγκη για τις νέες τεχνολογίες και θα πρέπει εμείς να διατυπώσουμε τα πρότυπα και την ομοθεσία που θα επιτρέψουν οι, οι αυτές, οι τεχνολογίες αυτές να βγουν στην αγορά γρήγορα έτσι ώστε για αυτή τη νέα τεχνολογία να υπάρξει μια ενιαία αγορά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε βιομηχανικό επίπεδο, γιατί είναι σαφές πως αυτές οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν πλεονεκτήματα και για τις μικρότερες επιχειρήσεις αλλά και τις μεγαλύτερες οι οποίες με τον τρόπο αυτό θα διατηρήσουν την αντιγωνιστικότητά τους και τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα στην παγκόσμια αγορά. Αυτά λοιπόν είναι κατά τη γνώμη μας σημαντικά. Και ίσως και ένα δεύτερο σημείο το οποίο δεν αναφέρθηκε εδώ, αλλά που έχει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο στην ανακοίνωσή μας, είναι η τυποποίηση και τα πρότυπα. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα τυποποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο λειτουργεί πολύ καλά. Όμως το σύστημα αυτό θα πρέπει παρόλα αυτά να βελτιωθεί έτσι ώστε να είναι τα πρότυπα χρήσιμα και στο μέλλον πρότυπα τα οποία θα μας κάνουν πιο ανταγωνιστικούς και που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε κοινωνικές προκλήσεις όπως η αλλαγή του κλίματος. Άρα λοιπόν αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο και θα ήθελα εκεί να ακούσω τις δικές σας απόψεις γιατί βέβαια στο χώρο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιδρά ε, με την ταχύτητα που ενδεχομένως θα έπρεπε να αντιδράσει Και το τρίτο στο οποίο αναφέρθηκα και το οποίο υπάρχει και αυτό στην ανακοίνωσή μας έχουν να κάνουμε την ενιαία αγορά. Δηλαδή, επιβολή της ενιαίας αγοράς. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε το πακέτο για τα προϊόντα και να οικοδομήσουμε την ενιαία αυτή αγορά παντού. Να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να έχουμε τις αρχές εποπτείας της αγοράς, ε, τις τελωνιακές αρχές για να έχουμε μια καλύτερη ενιαία αγορά, να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα με τα πλαστά ή παραποιημένα προϊόντα, τέτοιου είδους θέματα, τα οποία κατά τη γνώμη μου σχετίζονται απόλυτα και με τις εργασίες και την εντολή της δικής σας Επιτροπής και τα οποία φαντάζομαι ότι σας ενδιαφέρουν. Τα κάνω αυτά τα σχόλια γιατί πιστεύω πως οι προτάσεις που κάνετε εσείς είναι εξαιρετικές. Χαιρετίζουμε, επαναλαμβάνω, τις προτάσεις και τα σχόλια των συναδέλφων και σίγουρα υπάρχει περιθώριο για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις προτάσεις σας αυτές. Ίσως λοιπόν το θέμα αυτό του πώς η Επιτροπή Ενίας Αγοράς μπορεί να συνεισφέρει ε, χρήζει κάποιον ε, κάπως περισσότερη σκέψη. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια που είναι τόσο ενθαρρυντικά. Ο κύριος Κρότσμαν έχει το λόγο. Ακούσατε λοιπόν κάτι επιπλέον. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να είναι πολύ ευσύνεπτη η πρόταση και μετά λένε κάποιοι ότι πρέπει να προσθεθούν και οι τροπολογίες. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, εγώ είμαι ευγνώμων για όλα αυτά και γι' αυτό το λόγο είδα ε, τι ε, έχει ο κύριος Λάγκεν στην έκθεσή του. Υπάρχουν αυτά τα κοινωνικά θέματα. Ε, κοιτάξτε, εγώ είμαι ευγνώμων για όλα αυτά τα οποία είπατε και αν θέλετε όλα αυτά μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε ε, με τροπολογίε. Δεν υπάρχουν διαφορέ. Μόνο με την κυρία Κέπχαρτ έχουμε πάντα διαφορέ. Τέλο πάντων, εντάξει, δεν είναι και τόσο τραγικό. Ε, πάντως ε, στη τελική ανάλυση όλες, όλα αυτά καλύφθηκαν από την έκθεση Λάγκεν. Νομίζω λοιπόν ότι οι συνεργάτες μου έγραψαν ε, όλα αυτά που είπατε. Κοιτάξτε συνάλφε, δεν νομίζω ότι διαφωνούμε. Ε, ίσως ε, πρέπει να αφήσουμε κάποια θέματα και να συμπεριλάβουμε κάποια άλλα. Ε, μπορεί κανείς να ασκήσει κριτική, αν θέλει. Ευχαρίστως να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη μας. Γνωρίζετε λοιπόν ότι γνωρίζετε το χρονοδιάγραμμά μας. Η 1η Δεκεμβρίου είναι η καταληπτική ημερομιλία για την κατάθεση τροπολογιών και θα συζητήσουμε το θέμα στις 10 ε, Ιανουαρίου. Αυτά είχα να πω. Δεν νομίζω ότι ε, διαφωνεί κανείς εδώ από τους ε, συναδέλφους. Μικρή έτσι διαφωνία πάλι με την κυρία Γκέπχαρτ. Κατά τα άλλα... Είναι πολύ ενδιαφέρον ο συνάδελφος ε, κύριος Σβάπ, ε, ε, ο δικός σας ο εισηγητής κατέθεσε κάποιες τροπολογίες, μπορώ να τις δεχτώ, εντάξει όχι όλες και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το να δούμε τελικά πώς θα διεξαχθεί η ψηφοφορία, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις, αλλά θα πρέπει να αλλάξει λιγάκι το σύστημα έτσι ώστε να έχω και εγώ λίγο περισσότερο χώρο να γράψω περισσότερα πράγματα. Κοιτάξτε κύριε Κρόσες, ε, το θέμα είναι ότι πρέπει κανείς να είναι πολύ ψήνοπτος όπως ε, και όλοι μας. Ε, πρέπει λοιπόν να μπορέσετε να συμπεριλάβετε ακόμα περισσότερες προτάσεις μετά από τη συζήτηση που έγινε. Φοβάμαι ότι θα σας φορτώσουμε με δουλειά κατά και των Χριστουγέννων, αλλά είμαι και σίγουρος ότι δεν σας πειράζει. Ε, βλέπω λοιπόν ότι θα υπάρξει πολύ ζωντανή ανταλλαγή απόψεων στις συνεδρίες των συντονιστών. Πάμε τώρα στην επόμενη έκθεσή σας για τον τουρισμό. Εκεί θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων για το έγγραφο της Κομισιόν 30 Ιουνίου για ένα νέο πολιτικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Και έχουμε την κυρία Κόμη, την οποία και καλωσορίζω ως αντιπρόεδρο, η Χάιντι δεν είναι εδώ. Ο Κυριάκος είναι εδώ από τον Ελληνικό Τουρισμό, Οργανισμό Τουρισμού. Έχουμε εδώ την κυρία Τσαρντίνη. Έχουμε και εκπρόσωπο από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων. Ο κύριος Κρόιτσμαν έχει το λόγο. Ποια είναι παρακαλώ η αποψή σα για το θέμα του τουρισμού. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρο. Ομολογώ εξεπλάγει λίγο. Εγώ ε, πρόσφατα έκανα κάποιο τουρισμό στην Ρινανία Παλατινάτο, σε αυτό το κρατήδιο και διαπίστωσα πόσο δύσκολο είναι όταν ε, έχουμε αμπελώνες το πώ γίνεται διαφήμιση. Και είδα πόσο δύσκολο είναι στην Ανία Παλατινάτο να υπάρξει ενιαία διαφήμιση. Ο καθένα θέλει τη δικιά του κατ' επέκταση λοιπόν πόσο μάλλον στην Ευρώπη. Όλα αυτά με προβλημάτισαν και θέλω να σας πω τις σκέψεις μου. Καταρχήν αυτό το οποίο δεν φύγεται στο έγγραφο της ε, Κομισιόν είναι ο τουρισμός χωρίς σύνορα. Ο τουρισμός ε, αυτός ε, δεν αφορά μόνο τα άτομα με αναπηρία αλλά και τους πιο ηλικιωμένου. Αυτός λοιπόν ε, είναι ένας ελπιδοφόρος τουρισμός που πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε στην Ευρώπη. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Οφείλουμε να συνδυάσουμε τον τουρισμό με άλλες πολιτικές. Η δική μου εμπειρία είναι ότι ε, στη Γερμανία τουλάχιστον ο τουρισμός δεν αντιμετωπίζεται με οριζόντια προσέγγιση όμως μην ξεχνάμε τη σημασία του τουρισμού. Εκείνο που επίσης πρέπει να προσέξουμε είναι ότι στη Γερμανία τουλάχιστον, ε, δεν ξέρω τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, ε, δεν έχουμε εκπαιδευμένους, ε, εκπαιδευμένα στελέχη. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Εκείνο που χρειαζόμαστε επίσης είναι η βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων. Ε, την, ε, την, το αίσθημα της ευρωπαϊκής υπηκότητας ε, ε, μπορούμε και πρέπει το αίσθημα αυτό να τον ισχύσουμε οφείλουμε να δημιουργήσουμε τη βάση γνώσεων στον τουρισμό να επεκτείνουμε τη βάση αυτή να υπάρχει καλύτερη συνεργασία με συναδέλφους σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο να βελτιώσουμε το www.tourismeurope.gr να βελτιώσουμε αυτή την ε, πύλη γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν τοπικοί τοπικοί, δικτυακοί τόποι, διεθνείς, Εκεί είναι η ε, πύλη εισόδου και πρέπει να σκεφτούμε ίσως και να κάνουμε και κοινή διαφήμιση. Θα ήθελα λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρώπη μπορεί να διαφημιστεί γενικότερα στον κόσμο. Αυτό αφορά και τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Αυτές είναι έτσι κάποιες ε, ιδέες που ήθελα να αναφέρω για το θέμα του τουρισμού ε, εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ας ακούσουμε τους κοιόδης συγητές. Τι πρέπει να μπει κατά την απόψή τους ε, στην έκθεση του κυρίου ε, Κρόιτσμαν. Η κυρία Κόμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο τουρισμός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τον προστατεύσει, πρέπει να παραμείνει η Ευρώπη ο πρώτος παγκόσμιος προορισμός. Για να το καταφέρουμε θα πρέπει να κάνουμε προτάσεις που πηγαίνουν προς την κατεύθυνση που ανέφερε ο εισηγητής. Θεωρώ ότι η οικονομική κρίση δημιούργησε μια πτώση στις τουριστικές δραστηριότητες. Ο τουρισμός ε, όμως έχει μια ανάπτυξη 5,6% και με τάση να φτάσει και το 8%. Πρέπει να ξεπεράσουμε την εποχιακότητα, τον εποχιακό χαρακτήρα του τουρισμού για να αναπτυχθεί. Επίσης θα πρέπει να, να εναρμονιστούν τα τουριστικά συστήματα, δηλαδή να υπάρξει μια τυποποίηση για τα ξενοδοχεία, να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό σήμα ε, ποιότητας για τα ξενοδοχεία. Καλό είναι αυτό, αλλά να υπάρχουν και κάποια κριτήρια, κοινά κριτήρια, τα οποία θα χρησιμοποιούμε για να ταξινομήσουμε τα ξενοδοχεία. Ε, επίσης, θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή αναγνώριση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών, γιατί η αναγνώριση γίνεται τελείως διαφορετικά από κράτος σε κράτος ε, και τα, οι απαιτήσει από κράτος σε κράτος είναι τελείως διαφορετικές. Να βελτιωθούν οι σχέσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου με το σήμα ποιότητας, στην ε, έκθεση Αρίας είδαμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το σήμα που προστατεύει τα, τους χώρους που πληρούν κάποιες προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών. Αυτό να συνδυαστεί και με τον τουρισμό, να υπάρξει δηλαδή και στον τουρισμό. Να δημιουργηθεί επίσης α, μια, ένας λευκός κατάλογος για τους ε, tour operator. Ε, θετικά. Δηλαδή όχι μόνο μαυροπίνακες, ε, αλλά και ασπροπίνακε, α πούμε. Ένα αντίστοιχο σύστημα με το RAPEX. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή ένα κατάλογο έτσι, πληροφοριακό για τον καταναλωτή, ούτω ώστε ο καταναλωτή να γνωρίζει ποιοι είναι οι καλύτεροι tour operator στην αγορά. Αυτό να το συνδυάσουμε και με μια εναρμόνιση που το ζητούν οι tour operator, αλλά και οι υπόλοιποι τουριστικοί φορείς σε ό,τι αφορά την, το ΦΠΑ. Να εναρμονίσουμε το ΦΠΑ στον τουριστικό τομέα. Ευχαριστώ. Um, Το να προωθήσουμε την Ευρώπη ε, είναι μια πολύ καλή ιδέα, κύριε Κρόιτσμεν. Χρειαζόμαστε όμως να έχουμε μια πιο ε, ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον τουρισμό. Όλοι οι ενδιαφέρομενοι φορεί να εμπλακούν, ε, να λάβουμε υπόψη μας επίσης την επίπτωση του τουρισμού σε άλλες πολιτικές, στην προστασία των καταναλωτών, στο περιβάλλον, στις μεταφορές, στην ασφάλεια, ενεργητική και παθητική. Ένας τρόπος για να προωθήσουμε τον τουρισμό είναι μέσω των ωφελών που έχουν οι τουρίστες όταν ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Να δώσουμε στους πολίτες προσπελάσιμη, αξιόλο, ε, αξιόπιστη και αντικειμενική πληροφορία, καθώς και υποστήριξη σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά τους. Ε, να ενδυναμώσουμε την εικόνα μας στο εξωτερικό, να υπάρξει ανταλλαγή των καλών πρακτικών μεταξύ των ενδιαφερομένων. Θα πρέπει να επεκτείνουμε προγράμματα, όπως το δίκτυο ε, για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, το το, την πύλη για την ε, Ευρώπη ως ε, τουριστικό προορισμό και την ε, Ευρώπη ως τουριστικό προορισμό αριστείας. Η Κομισιόν όμως θα πρέπει να δώσει περισσότερα κονδύλια για τις τουριστικές πολιτικές. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε περισσότερα προϊόντα συγκεκριμένα σε νέες αναδυόμενες αγορές στη Βραζιλία, την Ινδία και την Κίνα εξειδικευμένα προϊόντα. Μετά την συνθήκη της Λισαβόνας, θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά για να διαμορφώσει τις τουριστικές πολιτικές. Θα πρέπει όχι απλώς να υιοθετούμε τις ίδιες προτάσεις, να έχουμε μια νέα στάση ε, και να μην εντοπίζουμε απλώς τα προβλήματα και τα διέξοδα. Κάτι στο οποίο ε, συμφωνώ με τον κύριο Κρόιτσμαν είναι στον ψηφιακό χώρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναγνωρίσει το δυναμικό και τις ευκαιρίες που μας προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ίντερνετ ε, στον τουριστικό κλάδο. Να βελτιώσουμε την πρόσβαση των καταναλωτών στην ψηφιακή αγορά μέσω της ολοκλήρωσης της ε, ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προωθήσουμε τον τουρισμό και μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών αλλά και από ξένους τουρίστες. Αυτά προς το παρόν. Συμφωνώ επίσης με αυτά που είπατε για την τυποποίηση και την κατάρτιση του τομέα του τουρισμού. Ευχαριστώ. Ο κ. Τριανταφυλλίδης. Ο κύριος De θα παρουσιάσει τις θέσεις μας. Είμαστε δύο σκιώδες, οπότε δίνω το λόγο στον κύριο De um, Uh, Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ αναγνωρίζω βεβαίως ότι υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα μέσω, που εξυπηρετούνται μέσω του τουριστικού κλάδου και βέβαια σε μια εποχή κρίσης καλό θα ήταν ε, να τα προωθήσουμε αλλά διάβασα με προσοχή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επειδή έχω και επιχειρηματική σκέψη πολλές φορές. Αναρωτιέμαι τι θα μας κοστίζει. Τι θα μας κοστίσει. Δηλαδή όλα αυτά τα συμβούλια, τα σήματα, ε, τα παρατηρητήρια, ε, το σήμα ε, ποιοτικού τουρισμού. Τι ακριβώς εννοείται και πόσα ευρώ θα κοστίσουν όλες αυτές οι προσπάθειες. Γιατί βέβαια δεν έχουν συμπληρωθεί αυτά στην πρόταση και φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι εξαιρετικά δαπανηροί. Επίσης, να σα πω πως υπάρχουν δύο είδη τουριστών. Υπάρχουν οι τουρίστες οι οποίοι θέλουν να τα δουν όλα ε, μέσα σε ένα πακέτο, ε, όπου τα τουριστικά πακέτα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, αλλά υπάρχουν και οι εξερευνητές, τουρίστες εξερευνητές. Βλέπω λοιπόν μια οικονομία με κεντρικό σχεδιασμό που έχει σκοπό να προγραμματίσει τα πάντα για τους τουριστές, εξ ε, αυτών και πιστεύω πως θα πρέπει να τους αφήσουμε, θα πρέπει να τους αφήσουμε και ένα πεδίο ε, ελευθερίας και επιλογής γιατί διαφορετικά αν ε, εφαρμόσουμε τα όσα έχουμε στην ε, ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χρειαζόμαστε χιλιάδες δημοσίους, δημοσίους υπαλλήλους. Ας προτιμήσουμε λοιπόν κάτι πιο ελαφρύ και χαλαρό. Τώρα, μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τουρίστες ε, που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης και επισκέπτεται την Ευρώπη. Η ανακοίνωσή σας ε, εστιάζει σε αυτούς και εκεί συμφωνώ με τη γενική φιλοσοφία, αλλά υπάρχει και ο ενδοευρωπαϊκός τουρισμός. Και νομίζω πως εμείς ε, θα συζητήσουμε και τις συντάξεις και τα όρια συνταξιοδότησης, αλλά μην ξεχνάτε ότι πριν από ορισμένα χρόνια, στα 55, οι συνταξιούχοι της Ευρώπης ζούσαν τη μισή τους ζωή σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος ε, και αυτά ως ε, σε ένα καθεστώς διαμονής. Άρα λοιπόν τώρα πια που αυξήθηκαν τα συνταξιδοτικά όρια, τι θα γίνει με αυτούς τους τουρίστες ας τους πούμε έτσι, ήταν ένα καλό μερίδιο της αγοράς το οποίο μάλλον θα εξαφανιστεί. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει ο σκιώδης μου και οι υπόλοιποι, οπότε ίσως θα μπορούσα εγώ να συνεισφέρω με κάποια σχόλια. Και δεν ξέρω βέβαια αν ο σκιώδης μου θα συμφωνήσει με τα σχόλιά μου, αλλά εγώ θα τα πω παρόλα αυτά. Θα επανέλθω στην πρόσφατη επίσκεψη που έκανα στην διάσκεψη για την ασφάλεια προϊόντων και να σας πω πως επισκέπτηκα και το ευρωπαϊκό περίπτερο όπου έγινε η διάσκεψη και αυτό το οποίο βρήκα πολύ ενδιαφέρον εκεί, πως στην έκθεση, κεντρικό έκθεμα ήταν ένα, ε, μια ταινία η οποία παρουσίασε μια ημέρα στην ζωή της Ευρώπης. Πολύ έξυπνα μονταρισμένο, ε, έδειχνε το τι γίνεται μέσα σε ένα σε διάφορες πόλεις και περιοχές της Ευρώπης. Άρα λοιπόν η ισχύ της Ευρώπης είναι αυτή τι πολιτιστική διαφορά που υπάρχει μεταξύ μας. Και νομίζω ότι αυτό αξίζει να επισκεφτεί κανείς. Εγώ δεν πιστεύω πως μπορούμε να προωθήσουμε την Ευρώπη ως ε, ε, εμπορικό σήμα. Έρχονται στην Ευρώπη γιατί τους αρέσουν αυτές οι διαφορές που μπορούν να επισκεφθούν, να δουν διαφορετικά τμήματα, με διαφορετικούς πολιτισμούς. Δεν νομίζω λοιπόν πως υπάρχει ένα image, ένα εμπορικό σήμα μία εικόνα της Ευρώπης που να μπορούμε ενιαία να προωθήσουμε. Νομίζω πως ε, πρέπει να το πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ συχνά τα επιχειρήματά σας, γιατί αν δείτε ε, τι κάνουμε εμείς και τα οποία ε, να είναι τουριστικού ενδιαφέροντος, νομίζω πως κάτι τέτοιο λείπει. Δεν βρήκα κάτι τέτοιο λοιπόν στο αρχείο μας. Τώρα η υπηρεσία, η οδηγία περί υπηρεσιών και το ότι ανοίξαμε τη διασύνοριακή αγορά για τις υπηρεσίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι μια φανταστική ευκαιρία για τις τουριστικές επιχειρήσεις είτε για να συνεργαστούν είτε για να έχουμε μεταφορά δεξιοτήτων και προϊόντων από χώρα σε χώρα με πιο εύκολο τρόπο. Αυτό δεν το αναφέρεται. Εμείς νομίζω το είχαμε βάλει στη γνωμοδότησή μας και σίγουρα και ο Κρότσμαν θα συμφωνήσει με αυτά που λέω. Δεύτερον, από τα όσα έχουμε κάνει, αλλά και από τα διάφορα αιτήματα και αναφορές που μας έχουν κατατεθεί, είναι η αμοιβή αναγνώριση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και κυρίως τις ε, τουριστικές δραστηριότητες, δηλαδή τουριστική οδηγή ξεναγή, που δεν έχουν το δικαίωμα να εργαστούν σε ξένες ε, χώρες, ε, μονιτέρ σκι και τέτοιου είδους επαγγέλματα. Άρα λοιπόν και αυτά θα πρέπει να αναφερθούν μια και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να διευκολύνουμε τη δράση αυτών των, αυτών του τύπου επιχειρήσεων. Τώρα για την ε, υπηρεσία που προσφέρεται για συνοριακά, ξέρουμε πως με την προώθηση των προτύπων ε, και για τις υπηρεσίες έχουμε καταφέρει κάτι το ιδιαίτερο και είναι πολύ σημαντικό και για την εφαρμογή της οδηγίας περιπηρεσιών από τα κράτη-μέλη. Αυτό λοιπόν που θέλετε να κάνουμε, αυτό το εμπορικό σήμα ποιοτικής τουριστικής επιχείρησης είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο για τα ξενοδοχεία, αλλά νομίζω πως θα έπρεπε εμείς να προωθήσουμε αυτές τις διατάξεις ε, με τους δείκτες ποιότητος που θα χορηγούνται σε τουριστικές επιχειρήσεις διασυνοριακά. περιβαλλοντολογικός τουρισμός, το αποτύπωμα του άνθρακα, ε, το κατά πόσο είναι φιλικό προς το περιβάλλον, φιλικός προς το περιβάλλον ο προορισμός προς τον οποίο ε, κινείστε. Επίσης, εγκαταστάσεις ασφάλειας και πόσο ασφαλείς είναι οι επιχειρήσει τι οποίε θα επισκεφτείτε. Έχετε οικογένεια, μικρά παιδιά και αγοράζετε πακέτο από το ίντερνετ. Θέλετε να ξέρετε εάν στην πισίνα του ξενοδοχείου που θα πάτε η πισίνα έχει φράχτη, προστατεύεται, έχει διασώστη και αν είστε ηλικιωμένο, θέλετε να δείτε τι υπηρεσίε σα προσφέρουν, παρουσία ιατρού κτλ. Η Επιτροπή μα βέβαια είναι γνωστή γιατί προωθεί το θέμα της ασφάλειας από πυρκαγιές στα ξενοδοχεία και νομίζω πως θα ήταν καλό να αναφερθούν όλες αυτές οι διαστάσεις γιατί είναι ένας τρόπος για να προωθήσουμε την Ευρώπη ως τουριστικό προορισμό. Ε, και εκεί θα λέμε ενιαία αγορά γιατί ναι, θα είναι ενιαία αγορά με την σκέψη πως θα είναι υψηλής ποιότητας οι υπηρεσίες που θα λαμβάνουν. Τώρα, για τις ε, κρατήσεις που γίνονται online και για τον τουρισμό online, αυτά είναι ζωτική σημασία για τον τουριστικό κλάδο. Όταν λέμε λοιπόν ενιαία αγορά, το πακέτο ε, για τα τουριστικά πακέτα και η οδηγία για τα τουριστικά πακέτα θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, καλά όλα αυτά. Χρειαζόμαστε και εδώ αρκετά στοιχεία και μπορούμε εμεί να προωθήσουμε ένα στεναρό βιώσιμο κλάδο και καλό θα ήταν όλα αυτά τα στοιχεία να τα συμπεριλάβουμε στις προτάσεις μας. Ωραία λοιπόν, αυτά. Κυρία Τζαρντίνη, δεν ήσασταν εδώ προηγουμένως. Προσπάθησα να σας καλωσορίσω, αλλά δεν ήσασταν. Αλλά θέλω να σας δώσω τώρα το λόγο να σχολιάσετε τα όσα ενδεχομένως ακούσατε από τους συγητές. Thank you. And sorry for being... Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι που αργήσαμε. Χαθήκαμε. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε και καλύτερη σηματοδότηση εδώ στο Κοινοβούλιο. Στείλτε επιστολή στο Προεδρείο. Σήμερα έχουμε συμμετάσχει σε τρεις ε, συναντήσεις και χαθήκαμε μόνο μία φορά, άρα το θεωρώ πολύ πετυχημένο. είναι πολύ ενδιαφέρον για μας να συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους συναντήσεις, το να ακούμε τις διάφορες προτάσεις που γίνονται σε αυτούς τους χώρους, γιατί κατά τη γνώμη μας η ανακοίνωσή μας είναι πολύ φιλόδοξη και πολύ πλήρης, με 21 δράσεις που προτείνονται. Αλλά βεβαίως υπάρχει χώρες ελεύθερους και για άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα πρέπει να εντάξουμε κάπως στο πλαίσιό μας παράλληλα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι νέε αρμοδιότητε υπό την συνθήκη τη Λισαβόνα και βέβαια να λάβουμε υπόψη πώ δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα. Παραδείγματο χάρη, εναρμόνιση, κατηγοριοποίηση ξενοδοχειακών καταλήμματων κτλ. Γιατί ξέρετε πω υπάρχουν και περιορισμοί δημοσιονομικοί. Για τη συζήτηση που έγινε σήμερα στις διάφορες συνεδριάσεις που πήγαμε, καταγράφουμε τις ε, ιδέες που ακούγονται και θα προσπαθήσουμε να τις λάβουμε υπόψη στο σχέδιο εφαρμογής που βρίσκεται στα σκαριά και το οποίο σχεδιάζεται με συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων είτε από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό κλάδο. Νομίζω πως μπορούμε να διευρύνουμε σε κάποιο βαθμό το υφιστάμενο σχέδιο και να λάβουμε υπόψη και τις ε, προτάσεις που καταθέσατε σήμερα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει κάποια παρανόηση για το ποιοι είναι οι στόχοι μας. Να είμαι λοιπόν πιο σαφής και να σας πω πως τα αποτελέσματα των όσων θα πετύχετε εσείς θα μας βοηθήσουν στο να επαναπροσανατολίσουμε τις προσπάθειές μας και κυρίως αναφέρομαι σε αυτό που αναφερθήκατε για τους συνταξιούχους που συνταξιοδοτούνται αργότερα από ό,τι στο παρελθόν. Θα μπορούσατε λοιπόν αυτά να τα χρησιμοποιήσετε σε κάποιες από τις δράσεις μας μέσω της πλατφόρμας που έχετε. Έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν περισσότερες ε, πληροφορίες, περισσότερες γνώσεις ε, για τις ε, τάσεις και να μπορούν να αποφασίσουν και το τι θα προσφέρουν για να ανταποκριθούν τις προκλήσεις. Θα λάβουμε λοιπόν υπόψη μας τις προτάσεις σας και σας ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας. Good. Well, Mr. would you like to perhaps uh, Κύριε Κρόιτσμαν, να απαντήσετε. Κοιτάξτε, αυτή η ε, ενιαία κατηγοριοποίηση των ξενοδοχείων. Ε, το είχα και εγώ στα δικά μου θέματα που ε, ήθελα να προβάλλω, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι αυτό γίνει και κάπου προαιρετικά. Πολύ σωστά το είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως. Βεβαίως ε, μπορεί κανεί να απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να του πει «Κοιτάξτε, εσεί να ταξινομήσετε τα ξενοδοχεία». Κάποιο πρέπει να κάνει ταξινόμηση και κάποιο πρέπει να την ελέγχει. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ήμουν λιγάκι επιφυλακτικό με το θέμα τη ταξινόμηση των ξενοδοχείων, γιατί σκέφτηκα ότι αν το ζητήσουμε αυτό, ε, καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως διαφορετικό από το να γίνει προαιρετικά και θα υπάρξουν ε, διαφορετικές απόψεις, ε, πολύ διαφορετικά τα πράγματα από το να πει κανείς αν θέλετε όλοι να μπείτε σε αυτήν την ενιαία, τον νέο τόπο του ίντερνετ θα πρέπει να προσφέρετε συγκεκριμένες πληροφορίες στους πελάτες που θα είναι φιλικές και σχετικά. Μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση ή αν θέλετε μπορούμε να πάμε στην Κομισιόν και να πούμε κάνε τα εσύ και να διαθέσει και τους πόρους. Όσον αφορά το θέμα της επικουρικότητας, ε, δίκιο έχετε ότι ε, δεν έχει νόημα άνθρωποι να έρχονται από την Ασία στην Ευρώπη και να μην ε, ξέρουν πού ακριβώς θα κατευθυνθούν. Θέλουν να πάνε στη Ρώμη, στο Παρίσι, στο Βερολίνο ή θέλουν να κάνουν σκι δεν έχει λοιπόν νόημα να τους πούμε ελάτε στην Ευρώπη, τελεία, χωρίς να διευκρινίζουμε απολύτως τίποτα. Εδώ πράγματι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την επικουρικότητα. Έλαβα υπόψη μου αυτά τα οποία ελέγχθησαν, τα άκουσα πολύ προσεκτικά. αν είχαμε περισσότερο χρόνο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε περισσότερο ε, και υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που έχουμε καταρτήσει. Η Κομισιόν όμως δεν ξέρω αν συμφωνεί 8 Δεκεμβρίου για, την, για το σχέδιο της χρηματοδότησης. Αν θέλετε μπορούμε το θέμα να το καθυστερήσουμε και μέχρι τον Ιανουάριο έτσι ώστε να ακούσουμε και άλλες απόψεις και μετά ε, θα γίνει ψηφοφορία ή δεν ξέρω ε, υπάρχει τεράστια πίεση ε, χρόνου. Εγώ έχω κάποιο χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρω αν είναι τεράστια η πίεση χρόνου. Εγώ θα προτιμούσα το σχέδιο αυτό να το συζητήσουμε μέχρι τον Ιανουάριο. Η ψηφοφορία προβλέπεται για τις 28 ε, Φεβρουαρίου. Ε, νομίζω λοιπόν ότι ε, αν συζητήσουμε και τον Ιανουάριο φτάνει ο χρόνος. Η αρμόδια επιτροπή, επιτροπή, επιτροπή χρόνια δεν να συνέρθει μέχρι τις 16 Μαρτίου. Αυτά ξέρουμε εμεί Ίσως ε, ξέρει κάτι η άλλη κυρία Τζορντίνη. Εμείς θα ψηφίσουμε λοιπόν στι 28 Φεβρουαρίου. Ε, εσείς έχετε λοιπόν ε, δύο εβδομάδες για να πάτε να τους πείσετε να συντάξουν τα σημεία μας στην τελική τους ε, γνωμοδότηση. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών είναι πολύ βολικός. Θα τον ειδοποιήσω ότι κάνουμε για τη δουλειά που κάνετε και ελπίζω να γίνουν δεχτέ οι μα στην γνωμοδότηση τη Επιτροπή Μεταφορών. Λοιπόν, αν δεν υπάρξει καμία αλλαγή, νομίζω ότι μπορούμε να δεχτούμε το χρονοδιάγραμμά σα. Δηλαδή, έχουμε μία προθεσμία. Μέχρι τότε πρέπει να σκεφτούμε τι ε, τροπολογίε. Το θέμα είναι αν μπορείτε να έχετε έτοιμη τη γνωμοδότησή σα λίγο νωρίτερα. Τώρα μιλάμε για την παρουσίαση της ε, γνωμοδότησης ε, στις 25 Ιανουαρίου. Έχουμε μόνο δύο μέρε για τις ε, τροπολογίε. Δεν νομίζω ότι αρκεί. Μήπω θα μπορούσατε να είστε έτοιμο ε, με την γνωμοδότησή σας ε, νωρίτερα, ούτω ώστε να ετοιμάσουμε και εμεί ωραιότατε τροπολογίες. Ε, θα μπορούσα να δώσω χρόνο στις μεταφραστικές υπηρεσίες και να είμαι έτοιμος το Δεκέμβριο. Αλλά το θέμα είναι τι νόημα έχει να δώσω την γνωμοδότησή μου λίγο πριν τα Χριστούγεννα, γιατί φεύγουν οι μεταφραστές. Ε, οπότε θα μπορούσα να στείλω το σχέδιο της εκθεσής μου μέσα Δεκεμβρίου. Μπορούμε λοιπόν να κρατήσουμε ως ημερομηνία ε, μέσα Δεκεμβρίου για την παρουσίαση της γνωμοδότησης για να έχουν χρόνο μεταφραστές. Οι υπόλοιπες ε, προθεσμίες, οι υπόλοιπες ημερομηνίες βολεύουν. Νωρίτερα λοιπόν από τις 25 Ιανουαρίου. Να την έχετε έτοιμη νωρίτερα λοιπόν από τις 25 Ιανουαρίου. Θα ήταν καλό αυτό. Τέλεια. Το... Η επόμενη ε, έκθεση δεν είναι του κυρίου Κρόιτσμαν, είναι του κυρίου Ντε Αφορά τα επαρκή ε, ασφαλή και βιώσιμα συνταξιδοτικά συστήματα στην Ευρώπη. Έχουμε τον κύριο Έγγελς. Ο κύριος Χανόκ δεν είναι εδώ. Η κυρία Γκέπχαρτ επίσης είναι παρούσα. Θα είναι σκιώδης. Ο κύριος Μάντος δεν είναι εδώ. Ε, τώρα, για αυτή τη γνωμοδότηση η, είμαι εγώ ο επίσημος σκιώδης ε, εισηγητής. Ο κύριος Ντεγιόγκ θα παρουσιάσει πρώτος τη γνωμοδότησή του και μετά οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομο θα είμαι. Νομίζω ότι δεν είναι μεγάλη γνωμοδότηση. Τέτοιες νομοδοτήσει δεν είναι μακροσκελής. Σας το έχω ξαναπεί ότι δεν θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να συζητήσουμε το θέμα των συντάξεων εδώ στη, για τις συντάξεις, γιατί η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή συζητάει αυτό το θέμα. Έχουμε όμως ένα-δύο στοιχεία που μπορούμε να συνεισφέρουμε κι εμείς ε, και αφορά τα δύο θέματα που μας απασχολούν εδώ, τα δικαιώματα των καταναλωτών και τα διασυνοριακά δικαιώματα που συνδέονται με την εσωτερική αγορά. Συμπεριέλαβα δύο βασικές αρχές, ούτως ώστε να καταλάβουν όλοι ότι γνωρίζουμε γενικώ αυτό το θέμα, ότι θα πρέπει να είναι επαρκή και βιώσιμε ε, και αηφόρε δηλαδή συντάξει, αλλά και αυτό που είπαν και άλλοι, ότι θα πρέπει να σεβαστούμε διάφορες συνθήκες ε, και επομένως ε, θα σεβαστούμε την αρχή της Επικουρικότητα. Για τα δικαιώματα των καταναλωτών είναι απλά τα πράγματα. Μιλάμε για τη διαφάνεια. Ο καταναλωτής πρέπει να είναι ενημερωμένος όταν αποφασίζει για τη σύνταξή του τις ατομικές, για τις ατομικές συντάξεις δηλαδή. Τα άλλα συστήματα είναι τα κρατικά ή τα υποχρεωτικά συστήματα συντάξεων. Αλλά τα μη υποχρεωτικά θα πρέπει να διέπονται από διαφάνεια. Να γνωρίζει κανείς τι περιμένει από τη σύνταξή του. Ε, κάποιες παράγραφοι, λοιπόν, λίγες παράγραφοι για τη διαφάνεια. Υπάρχει μια παράγραφος επίσης, θα το περιμένατε κύριε Πρόεδρε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εκείνοι που είναι μεμονωμένοι πάροχοι υπηρεσιών και που συχνά δεν έχουν τα λεφτά ούτε την πρόσβαση σε επαρκή ταξιδιωτικά συστήματα. Ε, χρήσιμο είναι στο τέλος της ζωής τους, όταν να σταματήσουν την εργασία τους, ε, ε, συχνά δουλεύουν ως ε, πάροχοι υπηρεσιών. Ε, θα πρέπει να στραφούμε προς τα κράτη-μέλη για να ενδυναμώσουν την πρόσβαση αυτών των κατηγοριών σε συνταξιδοτικά συστήματα. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό για τον καταναλωτή, αλλά αφορά και έχει σχέση με τα διασυνοριακά δικαιώματα. Αν κανείς έχει συνεισφέρει ε, σε συνταξιδοτικά συστήματα περισσότερα του ενός ε, κρατών μελών, δηλαδή, θα πρέπει να γνωρίσει ποια είναι τα δικαιώματά σου και επομένως να υπάρχει ε, ένα, ε, μια σύνδεση ε, μεταξύ των εθνικών συστημάτων, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχει σύνδεση των διαφόρων συστημάτων. είναι μια μακρόπνοη δουλειά, πρέπει να το αναφέρουμε. Πάμε τώρα στα διασυνοριακά δικαιώματα. Είναι η μεταφορά των συντάξεων. Αυτό είναι πάρα πολύ περίπλοκο θέμα έχει να κάνει και με τη φορολογική πολιτική. Αν έχει συνεισφέρει σε ένα κράτο ε, και δεν έχει φορολογηθεί εκεί όμω και αργότερα όταν φτάσει ε, στην εποχή τη σύνταξη, α, πώς μπορεί να μεταφέρεις ε, το ΣΥ, τη σύνταξή σου από το ένα κράτος ε, στο άλλο. Χρειάζεται ειδικό καθεστώς για να γίνει αυτό. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Επίσης, πώς υπολογίζονται τα δικαιώματα μέσα στα... Είναι θέμα των συνταξιωτικών ταμείων να υπολογίσουν το ύψος της σύνταξης που δικαιούται κανείς να μεταφέρει σε κάποιο άλλο, από ένα σύστημα σε ένα άλλο σύστημα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν προβλήματα με την οδηγία IORP, ιδίως ό,τι αφορά τους ορισμούς και κυρίως ε, τον ορισμό της διασυνοριακής δραστηριότητας. Στη χώρα μου, παραδείγματος χάρη την Ολλανδία, η κυβέρνηση θεωρεί ότι η διασυνοριακή δραστηριότητα ή μάλλον αν δουλεύει κανείς σε μια πολυεθνική με διάφορα παρατήματα μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το ίδιο ταξιδιωτικό ταμείο. Αλλά αυτό δεν θεωρείται διασυνοριακή δραστηριότητα. Σε άλλα κράτη-μέλη έχει σημασία που βρίσκεται η εταιρεία για να καθορίσουμε αν είναι ε, διασυνοριακή δραστηριότητα. Στην περίπτωση που ανέφερα, ε, είναι διασυνοριακή δραστηριότητα, γιατί η πολυεθνική που ανέφερα ε, δεν έχει την έντρα της στην Ολλανδία και αυτό οδηγεί σε συγχύσεις. Επίσης υπάρχουν πολλά εμπόδια για τις ασφαλίσεις και θα θέλαμε τις προτάσεις της Κομισιόν για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα πολλά θέματα για μια σελίδα, αλλά περιοριζόμαστε στις αρμοδιότητές μας. Ευχαριστώ κύριε Ντε Καλύψατε πολλά σημεία με συνοπτικό τρόπο. Δεδομένου και του περιορισμού της έκθεσης. Α, με προκαλέσατε με την IORP ως πρόεδρος Θέλω να σας μιλήσω ότι είναι το Ινστιτούτο για την σύνταξη, τις επαγγελματικές μάλλον συντάξεις. Όλοι θα γνωρίζετε τι είναι, εγώ δεν το ήξερα, τώρα το έμαθα. Ας συζητήσουμε λοιπόν και ας ακούσουμε πρώτα απ' όλα τον κύριο Έγγελ από τους κοιόδης συγητές. Σύντομα, Πρόεδρε. Αυτό που είπε ο κύριος Ντεγιόγκ δεν προσθέτει και πολλά καινοφανή. Ίσως ε, ένα φιλοσοφικό έτσι θέμα. Είχα την εντύπωση, διαβάζοντας την έκθεση, ότι εστιάζουμε στις, ε, στα επικουρικά συστήματα συντάξεων, στα, στις ιδιωτικέ συντάξεις επίσης. Τουλάχιστον στο γαλλικό κείμενο, διαβάζω το εξής. Στην παράγραφο 7 ότι μόνο οι υποχρεωτικές συντάξεις με βάση α, το σύστημα των επαγγελματικών συντάξεων είναι θεωρητικά μεταφερόμενες από κράτος σε κράτος. Θεωρητικά γίνεται αυτό. Στην πράξη δεν γίνεται. Δεν μπορεί να μεταφερθούν αυτά τα δικαιώματα. Θα ήθελα επίσης κάπου να βάλουμε μια προσθήκη σε κάποια παράγραφο που υπάρχει, μια νέα παράγραφο για να επισημάνουμε στην αρμόδια επιτροπή ότι πάντα, ότι ακόμα υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά τη μεταφορά δικαιωμάτων σε αυτό που λέμε στο Λουξεμβούργο, το νόμιμο σύστημα. Το νόμιμο ε, σύστημα που βασίζεται στις συνεισφορές και το οποίο είναι ανταποδοτικό. Σε καμία περίπτωση στην εσωτερική αγορά δεν μας ε, εξασφαλίζει μια σιγουριά ε, αυτό το σύστημα στο τέλος της επαγγελματικής μας ζωής, ειδικά όταν έχουμε δουλέψει σε διάφορα κράτη-μέλη. Κάπου θέλω να βάλουμε αυτή την ανησυχία. Εντάξει, άκουσα τα άλλα που είπε ο κ. De Όλα αυτά, τα υπόλοιπα μάλλον είναι σωστά, όλα είναι λογικά, αλλά παρακαλώ κάπου βάλτε και αυτό το θέμα. Κύριε, Πρόεδρε, ε, πρέπει να ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του συναδέλφου μου, ο οποίος βρίσκεται σε μια άλλη επιτροπή, όπου δυστυχώς και εκεί πρέπει να μιλήσει. Ως εκ τούτου μου παρέδωσε το κείμενο, ε, το οποίο θα διάβαζε και θα το διαβάσω κι εγώ, είναι στα γαλλικά. Εκτός μικροφώνιο, μιλήτρια. Παρό. Αναγνωρίζω λοιπόν πως πρόκειται μόνο για γνωμοδότηση και δεν είναι το σωστό πλαίσιο για να ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση για την συντάξη στην Ευρώπη. Αλλά χωρίς να ανοίγω το κουτί της Πανδώρας πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε κάτι πιο επιτακτικό και κρίμα που το κομμάτι που αναφέρεται στις ε, γενικές εκτιμήσεις είναι τόσο περιορισμένο. Φαντάζομαι πως ήθελα να το περιορίσει το ελάχιστο εισηγητής για να αφιερωθεί για τα στοιχεία που αναφέρονται περισσότερο, που μάλλον που είναι πολύ πιο σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Αλλά εάν περιοριστούμε στο να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία από την Πράσινη Βίβλο που μιλάει για συστήματα επαρκούς συνταξιοδότησης, τότε δεν διατυπώνουμε καμία γνώμη για τα συστήματα τα συνταξιδοτικά που επιθυμούμε να ισχύσουν για τους Ευρωπαίους συνταξιούχους. Παρόλο που αυτή τη στιγμή διατηρούν απλήρη ε, αρμοδιότητα λόγω της αρχής επικουρικότητας τα κρατημέλη στο θέμα της συντοξιοδότησης. Όμως στα πλαίσια της εντολής μας για την προστασία του καταναλωτή, όπως επίσης και για τις υπηρεσίες κοινή ωφέλεια, έχουμε το δικαίωμα να παρουσιάσουμε συστάσεις γενικής φύσης. Άρα λοιπόν, ε, τι σημαίνει σύστημα συνταξιδότησης κατά τη γνώμη μας. Καταρχήν πρέπει να είναι βιώσιμο, γιατί αν η χρηματοδότησή του δεν εξασφαλίζεται μακροπρόθεσμα, είναι οι πολίτες και κυρίως οι οικονομικά πιο ευάλωτοι, οι οποίοι θα πληρώσουν τον λογαριασμό. Όποιο λοιπόν σύστημα συντοξιδότης θέλει να φέρει το όνομα αυτό θα πρέπει να καλύπτει τις εξής ανάγκες, να εξασφαλίζει τα δικαιώματα για όλους και συντάξει οι οποίες θα επιτρέπουν στους συνταξιούχους να ζήσουν με αξιοπρέπεια. να μοιράζουν με ισότιμο τρόπο την προσπάθεια έτσι ώστε οι εισφορές να προέρχονται από όλα τα εισοδήματα λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές οικονομικές καταστάσεις ε, που έχει κάθε πολίτης και να υπάρχει και ένας βαθμός ευελιξίας έτσι ώστε σύμφωνα με την προσωπική πορεία του καθένα να μπορεί να κάνει την επιλογή που ταιριάζει στις ανάγκες του. Αυτή είναι λοιπόν η στόχη. Βιωσιμότητα, καθολικότητα, δικαιοσύνη και προσαρμοστικότητα. Για το υπόλοιπο του σχεδίου μονομοδότης, ο κύριος Ντεγιόμια έχει δίκιο υπογραμμίζει την ανεπάρκειά του στο μεταφορά των συνταξιδοτικών δικαιωμάτων από χώρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να άρει τα εμπόδια που ακόμα ε, αντίθετα στο σχέδιο γνωμαδότησης ε, εστιάζεται κυρίως ε, στον τρίτο πυλώνα που αφορά λίγους Ευρωπαίους και όπου η χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε ε, το πόσο ευάλωτο είναι γιατί τα συνταξιδοτικά ταμεία έχουν καταρρεύσει από τη μία μέρα στην άλλη, όπως επίσης ε, και οι επενδύσεις τους. Άρα λοιπόν έχουμε τις, ε, τα ατομικά συστήματα και καθεστώτα συνταξιοδότης όπου θα έπρεπε οι προτεραιότητες μας είναι η ορθή λειτουργία έτσι ώστε οι συντάξει των Ευρωπαίων πολιτών να εξασφαλίζονται γιατί από αυτά τα μία εξαρτώνται οι συντάξει τους και θέλουμε στην Ευρώπη στην οποία ζούμε να υπερισχύσει η αλληλεγγύη. Και πρέπει να σας πω πως αυτό είναι το κείμενο που μου έδωσε ο συνάδελφος και θα συμφωνήσω πλήρως με τα όσα γράφει. Ευχαριστώ. Πολύ κομψή η συνεισφορά του συναδέλφου σας και πολύ ωραία τα διαβάσατε. Νομίζω ότι είμαι ο τελευταίος σκιώδης ο οποίος βρίσκεται εδώ, άρα λοιπόν και εγώ πρέπει να σχολιάσω. Το θέμα είναι πως κάθε κράτος μέλος έχει τελείως διαφορετικά συστήματα συνταξιδοτικά και υπάρχουν εδώ θέματα και φορολογικής φύσης, αλλά και λειτουργίας των φορολογικών συστημάτων αυτών. Αυτά είναι ζωτική σημασία γιατί επηρεάζουν ε, για παράδειγμα τα κίντρα που δίδονται στην, ε, στις ε, συνεισφορές που πληρώνονται στα συνταξιδοτικά ταμεία, όπως επίσης και το τι κάνει κανείς να μετακινείται από χώρα σε χώρα. Έχετε δίκιο. Η ρύθμιση των καθεστώτων συνταξιδότηση και των σχετικών ταμείων είναι ελλειπής, αλλά ακόμα δεν έχουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που να ρυθμίζει τα συνταξιδοτικά ταμεία. Νομίζω πως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανερχόμενη ε, βέλτιστη πρακτική στο χώρο, αλλά φτάνει ως εκεί μόνο. Για την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νομίζω πως το θέμα των διασυνοριακών δικαιωμάτων πρέπει να συζητηθεί από εμάς, γιατί η κινητικότητα των ανθρώπων μας αφορά άμεσα. Έτσι έχουμε λοιπόν αμοιβή αναγνώριση δεξιοτήτων, διασυνοριακή κινητικότητα, και σε σχέση με αυτά, καλό είναι να παροτρύνουμε τους νέους νωρίς στην καριέρα τους, που είναι πιο κινητικοί και μετακινούνται από χώρα σε χώρα, να τους πούμε ότι κάνοντας αυτή την επιλογή καριέρας δεν θα βρεθούν σε δυσχερέστερη θέση ε, ε εν ώψη της σύνταξης σε σχέση τουλάχιστον με τα άτομα που δεν ε, μετακινούνται καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ξέρετε πως η σώρευση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από την αρχή της καριέρας σας έχει αποκτήσει όλο ένα και μεγαλύτερη αξία μεγαλύτερη αξία από ό,τι στο παρελθόν γιατί τα συνταξιδοτικά ταμεία πληρώνουν χαμηλέ συντάξει, γιατί τα συνταξιδοτικά ταμεία βρίσκονται όλα σε δυσκολίε λόγω τη αύξηση του προσδόκιμου ζωή και ότι υπάρχουν περισσότεροι συνταξιούχοι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτά τα ταμεία για πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Και βέβαια το προσδόκιμο ζωή εξακολουθεί να αυξάνεται. Άρα λοιπόν ο συνδυασμό αυτών των παραγόντων έχει κάνει τόσο δύσκολη την εξασφάλιση ε, των συντάξεων ε, των πολιτών. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε κάποια από αυτά τα θέματα και ο κύριος De βρήκε κάποια από αυτά γιατί νομίζω ότι συνδυάζονται με τα θέματα τα οποία ε, εμείς συζητάμε και στα οποία προσφέρουμε κάτι παραπάνω. Τέλος, έχουμε μια σημαντική πρόταση από την κυρία Γκέγγεν Κουίν. Αν μιλάμε για κατηγορίες ε, ατόμων που μετακινούνται, οι ερευνητέ στα πανεπιστήμια έχουν σκοπό τη μετακίνηση και τη μεταφορά γνώσεων και ψάχνουν τις καλύτερες ευκαιρίες για να μπορέσουν να μετακινηθούν και να χτίσουν την καριέρα τους. Ε, στο χώρο της Ευρωπαϊκής Έρευνας ελπίζουμε. Έχουμε λοιπόν την πρόταση της κυρίας Γκέγκεν Κουίν στην πρόταση της περί η Ένωση της Καινοτομίας, όπου θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν πειραματικά οι ερευνητέ, για να δούμε αν μπορούμε να στήσουμε ένα πανευρωπαϊκό ταμείο συνταξιοδότηση ερευνητών που θα επιτρέψουν σε όποιους θέλουν να κάνουν καριέρα στην έρευνα και στον πανεπιστημιακό χώρο να μην αντιμετωπίζουν ε, το μειονέκτημα ε, του ότι μετακινούνται από ίδρυμα σε ίδρυμα και μειώνεται με τον τρόπο αυτό η μελλοντική του σύνταξη. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν θα έπρεπε το πρόβλημα της συνταξιοδότησης να αποτελεί αντικίνητρο στη μετακίνηση ερευνητών και στη μεταφορά της γνώσης. Και εμεί, επειδή είμαστε Επιτροπή Ενιαίας Αγορά, νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τροπολογίε τέτοια φύσης θα ήταν πολύ χρήσιμες. Ωραία λοιπόν. Αυτά είχα να πω σκιώδη και. Σίγουρα ο κύριο Ντεγιόν θέλει να ακούσει την άποψη τη Κομίσιον. Έχουμε τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Φοβάμαι πως το όνομά σας δεν μπορώ να το προφέρω σωστά. Θέλετε να λάβετε το λόγο εκ μέρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντεγιόν για να κλείσει το θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα βέβαια θα λέω να ευχαριστήσω όλους σας ε, για την έκθεση και για τις παρεμβάσεις σας. Η πράσινη ε, βίβλος ξεκίνησε για να θίξει ακριβώς το θέμα της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής ε, για τις συντάξεις. πάρα πολύ ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό και ως εκ τούτου εμείς σχετίζουμε την έκθεση της Επιτροπής και της Επιτροπής αυτής Αυτή λοιπόν ε, η το πράσινο αυτό έγγραφο είναι μια ολιστική προσέγγιση απέναντι στις ε, συντάξεις όχι για ένα συγκεκριμένο στόχο αλλά για να μπορέσουμε να ε, δούμε τα πράγματα υπό ευρύτερο πρίσμα. Επ' αυτού νομίζω ότι σχολήσαν και οι συνεισηγητές. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω, ίσως ο συνάδελφός μου θέλει να προσθέσει κάτι, αλλιώς ε, μπορούμε και να κλείσουμε εδώ. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος και Ντιγιό, Ίσως θα έπρεπε να μιλήσουμε λιγάκι για το χρονοδιάγραμμα για να δώσουμε μια ε, τελική μορφή στην εκθεσία. Έχουμε δηλαδή το εξής. Θα ψηφίσουμε στις 26 Ιανουαρίου Καταληκτική ημερομηνία τροπολογιών 16 ε, Δεκεμβρίου, 12 η ώρα. Άρα δηλαδή θα μπορέσουμε έτσι να πάμε στην καθήλυνα αρμόδια επιτροπή που είναι η Επιτροπή Επασχόλησης. Ε, θέλετε να κάνετε κάποια σχόλια για να κλείσουμε το θέμα. Κοιτάξτε, θα ήθελα απλά να απαντήσω στις παρατηρήσεις που έγιναν. Και θέλω να πω ότι είχε δίκιο ο κύριος Ιωνοβάς με την έννοια ότι ε, υπάρχουν ε, κάποια πράγματα που λέγονται θεωρητικά ως εκ τούτου ε, δεν είναι και τόσο σημαντικά. Και εγώ ε, θα ήθελα να περιορίσω λιγάκι, μάλλον να εργαστώ μαζί για να διευρύνουμε το πλαίσιο. Όσον αφορά τώρα τις παρατηρήσεις που έγιναν μέσω της κυρίως Γκέπχατ, νομίζω ότι αυτά που άκουσα είναι η δικαιοσύνη ως αρχή, και εγώ βεβαίω ε, συμφωνώ και πρέπει να προσθεθεί, απλά δεν θα ήθελα να ανοίξω το κουτί της ε, Πανδώρας όπως ε, αναφέρθηκε και στην παρέμβασή της. Αν μπορεί κανείς να βρει κάποια ε, γενική διατύπωση, συμφωνώ, αλλά το να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας ε, και να ξεκινήσει μια, ξεκινήσει μια πολύ συγκεκριμένη κοβέντα για διάφορα θέματα, νομίζω ούτε εγώ το θέλω, ούτε και η Επιτροπή Απασχόλησης, που είναι κατά κύριο λόγο αρμόδια. πρέπει να σας πω ότι δεν κατάλαβα ακριβώς ε, αυτό που ελέγχεται ότι ε, στοχεύουμε κυρίως ε, στις συντάξεις του τρίτου πυλώνα. Βλέπετε εδώ υπάρχουν πάρα πολλά και για τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα. Ε, πάντως, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να περιμένουμε τις ε, τροπολογίες και να δούμε αν υπάρχει κάτι που μπορεί να αλλάξει. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, αυτά που είπατε εσείς ως εισηγητής σχετικά με την έρευνα ηχούν ε, ενδιαφέροντα. Σκέφτηκα τις πρακτικές επιπτώσεις που θα προεκυπταν αν υπήρχε η απέτηση ε, το να έχει κανείς αυτή τη στιγμή μία επαγγελματική ε, σύνταξη, σε ποια κατηγορία εμπίπτει και πώς σχετίζεται αυτή με την σύνταξή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με το γενικό στόχο, αλλά εδώ ε, το θέμα των συντάξεων είναι ένα ναρκοπαίδιο και πάρα πολλές πρακτικές εφαρμογές θα είναι δύσκολες. Ε, να δούμε λοιπόν τελικά πώς θα μπορέσουμε να τα συντάξουμε όλα αυτά, να δώσουμε μια γραπτή μορφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε την παρέμβαση της κυρία Χαμνόκ ε, μέσω της κυρίας Γκέπχαρτ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι σε αυτά που είπε η κυρία Γκέπχαρτ. Πάντως ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνατε για το θέμα αυτό και είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Τιγιόν ε, προσβλέπει στις ε, τροπολογίες σας. Θέλετε να προσθέσετε τίποτα άλλο. Όχι, δεν χρειάζεται. Πολύ ωραία λοιπόν. Απλά ήθελα να